Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο χρόνος τρέχει και έχουμε πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Έχουμε και μια κοινή συνεδρίαση με την ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ονομάζομαι Τσέσουαφ Σεκέρσκι και είμαι πρόεδρος τη Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξη. Και με ιδιαίτερα χαρά κηρύσω την έναρξη τη δημόσια αυτή ακρόαση και καλωσορίζω θερμά όλου ε, του συναδέλφου σε αυτή την κοινή, επαναλαμβάνω, συνεδρίαση των Επιτροπών Γεωργίας και Περιβάλλοντο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την ε, Λετωνική Προεδρία και τον Επίτροπο Άντριου Κάιτης για την αποδοχή της πρόσκλησης και την παρουσία τους στην σημερινή μας δημόσια κρόαση. Όπως γνωρίζετε, η δημόσια αυτή ακρόαση γίνεται στα πλαίσια της προετοιμασίας του νομοθετικού μας έργου, στα πλαίσια δύο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, για τις οποίε είναι συναρμόδιε οι Επιτροπέ Γεωργία και περιβάλλοντο. Γι' αυτό και έχουμε ορίσει και δύο συνεισηγητέ, την κυρία Τζούλη Μόη, εκ μέρου Επιτροπή Γεωργία, και την κυρία Ρενάτε Ζόμερ, εκ μέρου τη Επιτροπή περιβάλλοντο. Καλώ ορίζω και τι συνεισηγητριέ μα, τις μα και σε λίγο θα του δώσω και το λόγο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι τουλάχιστον το 2008, με την, ε, ότι από το 2008 με την ε, έγκριση του ψηφίσματος 3 Σεπτεμβρίου 2008 για, το, για την κλωνοποίηση των ζώων, ξεκίνησε από την Επιτροπή Γεωργίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, η προσπάθεια για υποβολή ειδικών προτάσεων για την κλωνοποίηση των ζώων που προορίζονται ε, σε παρασκευή τροφίμων. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, πολύ περίπλοκο και πολύπλευρο. Γι' αυτό και διοργανώνουμε αυτή την ακρόαση για μια ανοιχτή και επικοδομητική συζήτηση των διαφόρων πλευρών και πτυχών αυτού του εξαιρετικά δύσκολου, πολυσύνθετου και ευαίσθητου κοινωνικά θέματος. Η δημόσια μας ακρόαση θα χωριστεί σε τρία τμήματα. Σε ένα εισαγωγικό τμήμα που θα ακούσουμε υψηλόβαθμους θεσμικούς εκπροσώπους, εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων. Μετά στο πρώτο πάνελ θα έχουμε τον αντίκτυπο στην ε, αγροτοπιστιστική βιομηχανία και στην ευημερία των ζώων και το δεύτερο πάνελ με τις επιστημονικές και διδολογικές πτυχές ε, και τα θέματα του καταναλωτών. Και μετά από κάθε πάνελ θα έχουμε χρόνο για ερωταπαντήσεις. Θα δώσω τώρα το λόγο στον αξιότιμο συνάδελφο Τζοβάνι Λαβία, που είναι ο πρόεδρος, όπως γνωρίζετε, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και κατόπιν θα δώσω το λόγο και στους δύο, στις δύο συνεισηγήτριες. Παρακαλώ κύριε Λαβία, έχετε το λόγο. I uh, Σας ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σικέρσκι για τα εισαγωγικά του λόγια. Το θέμα της κλωνοποίησης των ζώων έχει επιμακρών ε, απασχολήσει την Επιτροπή μας, ε, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και ασφάλεια των Τροφίμων, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, ε, από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία συνδιαλλαγής ε, σε σχέση με τα πρώτη πρόταση περί νέων τροφίμων το 2011, η οποία απέτυχε ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν, υπήρχε συμφωνία για τις διατάξεις για την κλωνοποίηση. Έκτοτε η Επιτροπή Περιβάλλοντος επανειλημμένα ζήτησε από την Κομισιόν να κάνει νέα πρόταση για την κλωνοποίηση χωριστή από αυτήν για τα νέα τρόφιμα που θα βασίζεται στη τελευταία προσφορά του Συμβουλίου επί της πρότασης συνδιαλλαγής. Οι προτάσεις της Κομισιόν της 18 Δεκεμβρίου 2013 επιτέλους απέδωσαν ε, απαγόρευση της κλωνοποίησης για στόχους ε, κτηνοτροφίας στην Ένωση, την εισαγωγή ζώων κλωνοποιημένων και την τοποθέτηση στην αγορά, την εμπορία τροφίμων από ε, κλόνους ζώων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ε, συγκεκριμένε διατάξει για την ανιχνευσιμότητα ή για την ετικετοθεσία. Ούτε περιλαμβάνονται διατάξει για την ανίχνευση ε, αναπαραγωγικού υλικού από κλόνου σε θέματα τα οποία ανέκαθεν θεωρούσε το Κοινοβούλιο πολύ σημαντικά. Γι' αυτό είμαι πολύ ευτυχή που αυτή η κοινή ακρόαση γίνεται σήμερα και διότι ο Επίτροπο Ανδρικάητη και Εξ ονόματος της ε, Προεδρίας, ο κύριος Σταλμέιστερς ε, της ε, Λετωνικής Προεδρίας δέχθηκαν να είναι σήμερα μαζί μας, μαζί με έξι διακεκριμένους εμπειρογνώμονες, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, ώστε να φωτίσουμε όλες τις πτυχές της κλωνοποίησης ζώων για στόχους εκτινοτροφίας, εν ώψη των επομένων βημάτων της νομοθετικής διαδικασίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και να ακούσουμε τώρα τις δύο συνεισηγητριές μας. Πρώτα, την κυρία Μόη, την εισηγήτρια της Επιτροπής Γεωργίας. Παρακαλώ κυρία Μόη, έχετε το λόγο χρόνου φίδου όμως. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ στην πρώτη συζήτηση αυτού του θέματος που είναι τόσο σημαντικό και που μας αφορά όλους. Το θέμα της κλωνοποίησης των ζώων είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση της κλωνοποίησης και των προϊόντων που προκύπτουν από αυτή όλων των πιθανών επιπτώσεων για την υγεία των συμπολιτών μας. Σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο έργο, γιατί θα πρέπει να αποφασίσουμε ένα κομμάτι του μέλλοντός μας, ε, το μέλλον της διατροφής μας, των συνηθιών μας και της κοινωνίας μας της, ίδια, Άρα λοιπόν ε, περιμένω τις απόψεις όλων σας, αλλά θα ήθελα να σταθώ και να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένες σκέψεις που για μένα είναι σημαντικές και για τις οποίες, από τις οποίες μάλλον θα ήθελα να ξεκινήσω την ανάλυση. Ε, υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα καταρχήν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει κοινή γραμμή. Αυτό το αποδεικνύει η αποτυχημένη συμφωνία του 2011 που σχετιζόταν με τα νέα τρόφιμα. Ακριβώ λόγω τη υπερίληψη τροφίμων που προκύπτουν από κλωνοποιημένα ζώα, επί τη οποία ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάστηκε να επανέλθει στα τέλη του 2013 με νέε νομοθετικέ προτάσει ώστε να αναζητήσει λύσει. Θα πρέπει να πω ότι η πρόταση τη Κομισιόν σε αυτή την πτυχή περιλαμβάνουν διάφορες αποδεκτές θέσεις επί των οποίων θα μπορέσουμε να βασιστούμε ώστε να ξεκινήσουμε την εργασία μας. Αναλύοντας αυτή τη νέα ε, πρόταση ε, διαπιστώνουμε ότι εξακολουθεί να υφίσταται μεγάλη ε, επιστημονική αβεβαιότητα. Όχι μόνο για την υγεία των ζώων, αλλά και για τις πιθανές και μη εύκολα διακρίσιμες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κατανάλωση τέτοιων προϊόντων από τον άνθρωπο και για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες. Στην αξιολόγηση της ΕΦΣΑ βρήκα διάφορες αμφιβολίες και αναλύοντας και διάφορες άλλες επίσημες μελέτες διαπίστωσα πως υπάρχουν πολλές ελλείψεις και που οφείλονται στην έλλειψη των ε, επιστημονικών ερευνών. Δεν υπάρχει ας πούμε βεβαιότητα για το ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή της, ε, ε επιλογή των ζώων. Τα κριτήρια επιλογής του είδους θα πρέπει να σεβαστούν αυτά που ισχύουν και στη φύση, γιατί διαφορετικά μπορεί να υπάρξει ο κίνδυνος διαφορετική επιλογής που είναι καρπός άλλων τεχνικών που θα μπορούσε να οθήσει στο να ερευνήσουμε τις επιπτώσεις με μεγάλη όμως ακρίβεια. Στην σύνταξη αυτή τη έκθεση, μαζί με την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και τη υγεία του, θα ήθελα να προσθέσω πω ανάμεσα στι προτεραιότητέ μα θα πρέπει να ε, ε, δώσουμε μεγάλη προσοχή και στην εξέταση τη κατάσταση των ζώων που ήδη ορίζονται ω ε, όντα που έχουν συνέστηση ε, από τη συνθήκη της Λισαβόνας έτσι ορίζονται. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε καμιά από αυτές τις διαστάσεις και τις ε, πραγματικότητες γιατί η ευημερία των ζώων θα πρέπει να είναι εγγυημένη όπως και η ασφάλεια των πολιτών και καταναλωτών της Ευρώπης. Και τα πράγματα αυτά τα δύο θα πρέπει να συμβαδίσουν απαραίτητο πρώτη συνάντηση για αυτό το θέμα με τεράστιες ευθύνες, ωστόσο είμαι βεβαία ότι σε συνεργασία με την συνάδελφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, τους κοιόδης εισηγητές και όλους εσάς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο έργο μας προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Περιμένω λοιπόν ώστε να ακούσω τα όσα θα μας πούν οι εμπειρογνώμονες που είμαι βεβαία να μας δώσουν πολλές λαβές επί των οποίων να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ ευχαριστώ κύριε Ζόμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ καλωσορίζω όλους τους συναδέλφους. Καλώς ήρθατε κι εσείς ε, κύριε Επιτροπέ και βεβαίως ε, Οπωσδήποτε ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε καλά και με τους δύο συνεισηγητές και μπορώ να σας πω πως και εγώ χαίρομαι και αναμένω τη σημερινή ακρόαση με μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι ε, οι οποίοι ίσως να μην είναι τόσο εξοικειωμένοι με το θέμα. Ε, το 2008 στην προπροηγούμενη θητεία ε, είχαμε ασχοληθεί με το θέμα του ε, της ε, κλωνοποίησης και μας απασχολεί και πάλι και μας απασχολεί γιατί ξέρουμε πως είναι βεβαίως πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να υπάρξει νομίζω μια περαιτέρω ρυθμίση αυτού του θέματος γιατί έχει φτάσει η στιγμή να υπάρξει. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά ήταν σχετικά ενωμένο. Δεν ε, ενθουσιάστηκε τότε με την ιδέα να έχουμε κλωνοποιημένα ζώα ή αναπαραγωγικό υλικό ή απογόνους τους ε, στην Ευρώπη και τώρα θα δούμε τι θα αποφασίσει αυτή την φορά. Υπάρχουν διάφορα θέματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν, προστασία των ζώων, των καταναλωτών, ε, ηθικής όπως το λέμε, και βεβαίως και το θέμα της γεωργίας. Ε, χρειάζεται πράγματι κτηνοτροφία, κλωνοποίηση για να είναι ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά. Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν σήμερα. Ελπίζω να έχουμε λοιπόν μια ενδιαφέρουσα ακρόαση. Και εύχομαι καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Με ιδιαίτερη χαρά θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γιούρι Σταλμάισταρς, που είναι ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος ε, της Λετωνίας ε, για να μας παρουσιάσει τις απόψεις ε, της Λετωνικής Προεδρίας. Παρακαλώ κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο. Κύριοι Πρόεδρε των Επιτροπών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, κελαβία και Λαβία, κύριε Επίτροπε Ανδριοκάητης, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ και καλεσμένοι, χαίρομαι ιδιαίτερος για την ευκαιρία που μου δίνετε να σα παρουσιάσω τις θέσεις Λετωνική Προεδρία σε αυτή τη δημόσια ακρόαση και κοινή συνεδρία των δύο επιτροπών γεωργία και Περιβάλλοντος για να σας παρουσιάσω και τις θέσεις του Συμβουλίου στα θέματα της κλωνοποίησης. Όπως και οι προλαλήσαντες, θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω με λίγα λόγια για το ιστορικό υπόβαθρο αυτής της πρότασης. Όπως ξέρετε, η πολιτική κλωνοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι μακροχρόνια και χαρακτηρίζεται από περίπλοκες θεσμικές συζητήσεις και μάλιστα επανήρθε στο πολιτικό, πρόβλημα μετά, στο πολιτικό πρόγραμμα μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις για τα νέα τρόφιμα το 2011. Ο βασικός λόγος αποτυχίας ήταν το θέμα των τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα ή από γόνους τους. Θέλουμε μια ισορροπημένη λύση, εύχρηστη, για να ικανοποιεί τις φιλοδοξίες ε, όλων των ενδιαφερομένων μερών, κάτι που δεν κατέστη δυνατό μέχρι τώρα έχουμε την ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπει ότι θα πρέπει να δίνεται προηγούμενη άδεια ε, εμπορευματοποίηση για τρόφιμα κλωνοποιημένα ζώα, κάτι, αλλά δεν απαγορεύεται η, κλωνοποίηση, η τεχνική κλωνοποίηση. Και όπως είπα το 2011 να βάγισαν οι διαπραγματεύσεις ε, στα νέα τρόφιμα. Είναι σημαντικό όμως ε, να αποφύγουμε στο μέλλον τα λάθη του παρελθόντος και να σημειώσουμε πρόοδο. Είναι σημαντική λοιπόν η συνεργασία του Συμβουλίου με το Κοινοβούλιο για τα νέα τρόφιμα και μάλιστα φαίνεται ότι η συνεργασία αυτή θα οδηγήσει σε ένα αίσιο πέρας. Με τα νέα τρόφιμα θέλουμε πρόσβαση νέων καινοτόμων προϊόντων στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας υψηλέ προδιαγραφές υγεία. Οι άλλε δύο προτάσεις για την κλωνοποίηση απαγορεύουν τις ε, ε, τεχνικές κλωνοποίησης ε, για τα ζώα εκτροφής, τα εισαγόμενα κλωπημένα ζώα και τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα. Και υπάρχουν και κάποιες ε, δεοντολογικές πτυχές στο θέμα της κλωνοποίησης. Τώρα, ποια είναι η προσέγγιση του Συμβουλίου. Για να αντιληφθείτε και πώς βλέπει ε, τα θέματα αυτά το Συμβούλιο. Είναι γνωστό ότι το Συμβούλιο πιστεύει ότι η κλωνοποίηση θα πρέπει να τύχει ξεχωριστή αντιμετώπιση από την πρόταση για τα νέα τρόφιμα. Γιατί η νομοθεσία για τα νέα τρόφιμα προβλέπει σταθερέ βάσει για την καινοτομία στην Ευρώπη και δεν θα πρέπει να συνδέεται με το θέμα τη κλωνοποίηση. Η Λεπτονική Προεδρία θα υποστηρίξει αυτή τη θέση. Επίση, θα ήθελα επ' ευκαιρία να καλέσω του ενδιαφερόμενου ε, στη διαπραγμάτευση να έχουν υπόψη αυτό το θέμα και να μην χάσουν την ευκαιρία να συμφωνήσουν με βασικά θέματα των νέων τροφίμων, όπως είναι η κεντρική διαδικασία αδειοδότησης, νομικός ορισμός των ανοηλικών και ειδικά μέτρα για τα παραδοσιακά τρόφιμα από τις τρίτες χώρες. Έτσι θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να έχουν μια ευρή επιλογή τροφίμων, αλλά σε ένα ασφαλές περιβάλλον και για την αγροπιστική βιομηχανία με υψηλές ε, προδιαγραφές υγείας. Σε ό,τι αφορά τι εργασίες του Συμβουλίου για την κλωνοποίηση, γίνεται προσεκτική τεχνική εξέταση της πρότασης ε, στο Συμβούλιο και γνωρίζετε όλοι πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα της κλωνοποίησης για τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα τώρα να σας, παρουσιάσω, να σας παρουσιάσω μερικά από τα βασικά στοιχεία της συζήτησης στο Συμβούλιο. Καταρχήν, επιλογή του νομικού μέσου, το πεδίο εμβέλειας των προτινόμενων μέτρων, η συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες και οι διατάξεις για τον έλεγχο. Ε, το Συμβούλιο θέλει ε, να βρει λύσεις με στέρεες νομικές βάσεις που ε, θα στηρίζονται στην, επιλογή, στην μελέτη επιπτώσεων, θα είναι εφαρμοστές, θα είναι παραπλανητικές για τους καταναλωτές και θα τηρούν τις διεθνείς μας εμπορικές υποχρεώσεις. Με όλα αυτά τα κριτήρια κατά νου και δεδομένης της ευαισθησίας του θέματος, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε μια ισορροπημένη συμβαστική λύση, ρεαλιστική, τεχνικώς εφικτή, που θα περιλαμβάνει και το θέμα της συχνηλασιμότητας και της ετικετοθεσίας για τα προϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα. Φυσικά παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το έργο του Συμβουλίου και ευελπιστώ ότι και τα δύο σκέλη της νομοθετικής αρχής θα καταλήξουν σε μια αποδεκτή λύση για αυτό το ευαίσθητο ζήτημα της κλωνοποίησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη για την παρουσίαση της ε, θέσης του Συμβουλίου και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο τον κύριο Άντριο Καϊτής για να μας παρουσιάσει την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Dear committee members. Αγαπητοί συμπρόεδροι, μέλη της Επιτροπής, συζητητές, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρόσκληση αυτή συνεκτή συνεδρίαση των επιτροπών σας και για το ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τις δύο προτάσεις της Κομισιόν για την κλωνοποίηση. Θα θυμάστε ότι ευθύθηκαν το Δεκέμβριο του 2013 επί προηγούμενης Κομισιόν. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω παρουσιάζοντας το περιεχόμενο των δύο αυτών προτάσεων. Η πρώτη πρόταση αφορά την αναστολή της κλωνοποίησης των ζώων. Έτσι θα απαγορευτεί η κλωνοποίηση βοηδών, χείρων, προβάτων, εγώ προβάτων και αλόγων και της ε, θέσης εμπορία κλωνοποιημένων ζώων και εμβρίων. Η δεύτερη πρόταση αφορά την ε, αναστολή της θέσης εμπορία κρέατος κλωνοποιημένων ζώων καθώς και ε, γαλακτοκομικών προϊόντων από κλωνοποιημένα ζώα. Η πρώτη πρόταση αφορά την ε, τεχνική της κλωνοποίησης και τα ίδια τα ζώα, ενώ η δεύτερη πρόταση αφορά το τα τρόφιμα από τους οργανισμούς αυτούς. Μετά από πέντε χρόνια η Κομισιόν θα κάνει μια τεχνολογική και επιστημονική εξέταση του ζητήματος καθώς και ζητήματα που αφορούν την ε, ευζοία των ζώων αλλά και ζητήματα ηθικής. Μετά θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το γεγονός πως ε, έρχομαι στην Επιτροπή Γεωργίας και Ασφάλειας Τροφίμων και Καταναλωτών δείχνει πως ε, έχουμε ένα ζήτημα περίπλοκο και πολύπλευρο. Είμαι αισιόδοξο ότι θα καταφέρουμε τελικά να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση όπως καταλήξαμε και για τους γενετικά τροποποιημένους ε, οργανισμούς. Ήταν αντικείμενο κανονισμού το 2011 και παρά τις προσπάθειες της Ουγγρικής ε, Προεδρίας απέτυχε η συνδιαλλαγή μετά από παραπάνω από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων. Κατόπιν λοιπόν η Κομισιόν σκέφτηκε τα ζητήματα αυτά και κατέληξε σε μια νέα νομοθετική πρόταση. Ως αποτέλεσμα αυτού η Κομισιόν προετοίμασε δύο ξεχωριστές πρώτης και αποσυνέδεσε την κλωνοποίηση από τα καινοτόμα τρόφιμα. Και αυτές είναι οι προτάσεις τις οποίες συζητάμε σήμερα. Εξέτασα, τις εξέτασα προσεκτικά και τώρα ήρθα να ακούσω τις απόψεις σας. Καταλαβαίνω πως τα ζητήματα αυτά είναι περίπλοκα και πρέπει να εξετάσουμε όλες τις πτυχές τους. Την ευζοία των ζώων, σεβασμό της γενετικής ποικιλία καινοτομία και έρευνα και βεβαίως να λαμβάνουμε σωστές αποφάσεις σημαίνει πως θα πρέπει να σεβαστούμε και τις ευαισθησίες και τα επιστημονικά δεδομένα. Όσον αφορά δε την ε, ασφάλεια των τροφίμων ε, δεν τίθεται ζήτημα τέτοιου κινδύνου. Όσον αφορά την ευζοία των ζώων, γεγονό είναι πως όλα τα ζώα τα οποία μπλέκονται στην κλωνοποίηση ε, υποφέρουν και οι κλόνοι και οι παρένθετες μητέρες. Οπότε δεν είναι δυνατόν να μεταχειριζόμαστε τα ζώα σαν να ήταν αντικείμενα. Αυτό φαίνεται άλλωστε και στο ότι η συνθήκη αναφέρει πως τα ζώα είναι νοήμωνα όντα. Και η εξολόγηση αντικτύπου αναφέρει πως ε, η κλωνοποίηση δεν είναι μία από τις καινοτόμες μεθόδους που χρειαζόμαστε, καθώς δημιουργεί και προκαλεί πόνο στα ζώα. Κάποιες τρίτες χώρες όμως έχουν κάνει μια διαφορετική επιλογή και έτσι ερχόμαστε στο θέμα των απογόνων κλώνων. Όπως ξέρετε εισάγουμε σπέρμα από κλωνοποιημένα ζώα για τη γονιμοποίηση ζώων στην Ευρώπη. Τα ζώα που γονιμοποιούνται έτσι έχουν τις ίδιες ε, συνθήκες εκτροφής όπως αυτά τα οποία γονιμοποιούνται με συμβατικό σπέρμα. Τίθεται λοιπόν ένα ζήτημα σήμανσης και εδώ πέρα δεν συμφωνείτε με την άποψη της Κομισιόν. Η εξολόγηση αντικτύπου για την σήμανση έδειξε πως η σήμανση για τα τέκνα και τους απογόνους ήταν περίπλοκη και ε, βεβαίως κοστίζει. Γι' αυτό αποφασίσαμε να μην την εφαρμόσουμε όμως, οπωσδήποτε θα εξετάσουμε το ζήτημα οι υπηρεσίες κομισιών έχουν ξεκινήσει μια μελέτη για, την, το εφικτό και τον πιθανό αντίκτυπο της σήμανσης ε, κλώνων και απογόνων. Η μελέτη θα είναι έτοιμη την Άνοιξη και ελπίζω έτσι να διαφωτιστούμε ως προς το θέμα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας. Και καλό είναι να ακούσουμε όλες τις επιλογές ε, για να προχωρήσουμε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Οπότε ολοκληρώσαμε το εισαγωγικό τμήμα της δημόσιας ακρόασης, ε, δηλαδή την παρουσίαση των εκπροσώπων θεσμικών οργάνων και θα περάσουμε στο πρώτο πάνελ. Ε, που θα μας παρουσιάσει θέματα που ενδιαφέρουν κυρίως στην Επιτροπή Γεωργίας. Αφορά προτάσεις ε, για την εκτροφή, την κτηνοτροφία των ζώων και την, ε, τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Θα δώσω το λόγο για σύντομες παρουσιάσεις στους καλεσμένους μας, εμπειρογνώμονες. Και πρώτα θα δώσω το λόγο στην ε, εισηγήτρια της Επιτροπής Γεωργίας, την κυρία Μόη. Ε, ehm, ε, ναι, εμείς στην Επιτροπή Άγκρη θα θέλαμε να αφήσουμε το λόγο σε κάποιους τεχνικούς για αυτό το θέμα, γιατί θεωρούμε ότι το πρόβλημα της υγείας και της ευημερίας των ζώων είναι σημαντικό. Όπως λέει και η συνθήκη της Λισαβόνα στο άρθρο 13 πρόκειται για ε, όντα με, ε, που, που αισθάνονται, που νιώθουν. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πόσο μπορεί να αποφέρουν τα ζώα μέσω αυτών των τεχνικών. Γι' αυτό και θα θέλαμε να ακούσουμε τώρα τους εμπειρογνώμονες που βρίσκονται σήμερα εδώ. Bardzo dziękuję. Oddam panu θα δώσω τώρα το λόγο στον πρώτο μας ε, καλεγρισμένο, τον κύριο Γιάννου Βένεμαν, για την πρώτη παρουσίαση. Είναι διευθυντής του Ευρωπαϊκού Φόρουμ ε, Εκτροφέων. Και θα του δώσω το λόγο για 10 λεπτά. Ο κύριος Βένεμαν είναι, αρμόδι, εμπειρογνώμονος και για θέματα αναπαραγωγής ζώων από το Πανεπιστήμιο του Βάγκενιγκεν και ήταν ε, επικεφαλής πολλών τμήματων του Ολλανδικού Υπουργείου Γεωργίας και επίσης σύμβουλος στον ημιδημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θα δώσω το λόγο στον πρώτο μας εμπειρογνώμονα λοιπόν, τον κύριο Βένεμαν για την παρουσίασή του. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Βένεμαν. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην πολύ σημαντική αυτή συνεδρίαση. Χαιρόμαστε που έχουμε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί σας. Πριν περάσω το θέμα θα ήθελα να εξηγήσω κάποια πράγματα για το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κτηνοτρόφων. Είμαστε μια ένωση του κτηνοτροφικού τομέα στην Ευρώπη τα μέλη μας είναι ιδιωτικές ενώσεις ε, του κτηνοτροφικού τομέα, αρκετοί συνεταιρισμοί κτηνοτρόφων, έχουμε σχεδόν 30 μέλη στην Ευρώπη. Ασχολούμαστε με όλα τα παραγωγικά ζώα, μυρικαστικά, πουλερικά, ηχθειοκαλλιέργεια, αλλά βεβαίως όσον αφορά την κλωνοποίηση μιλάμε κυρίως για χείρους και μυρικαστικά και μιλάμε για ε, κτηνοτροφία και ε, αναπαραγωγή. Βεβαίως ε, η κλωνοποίηση δεν είναι κτηνοτροφία, είναι αναπαραγωγή, αλλά επηρεάζει οπωσδήποτε την κτηνοτροφία. Στόχος μας είναι λοιπόν να προωθήσουμε τα συμφέροντα των μελών μας ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Κομισιόν, σε σχέση με διάφορα ζητήματα για την τεχνική νομοθεσία, την ευζοία των ζώων, αλλά εμπλεκόμαστε και σε ερευνητικά ζητήματα. Προσπαθούμε να συνεισφέρουμε και στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 όπως έγινε και το 2014-2015 και βεβαίως ε, προωθούμε τις ευρωπαϊκές ε, ερευνητικές ε, δραστηριότητες. Για την κλωνοποίηση έχω μόνο μία διαφάνεια. Λοιπόν, κλωνοποίηση ζώων την λέω πρόταση κλωνοποίησης και την άλλη πρόταση την λέω πρόταση εμπορίας. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, η πρόταση για την κλωνοποίηση εξηγήθηκε ήδη, απαγορεύει την κλωνοποίηση των ζώων απαγορεύεται η εισαγωγή εμβρίων κλώνων και κλώνων ζώων, αλλά προσέξτε αυτό δεν σημαίνει ε, έμβρια κλώνων, δεν σημαίνει ε, δεν σημαίνει ε, απογόνους των κλώνων. Μιλάμε απλά για το κλωνοποιημένο ζώο το οποίο είναι έμβριο, αλλά όχι για τα έμβρια αυτού. Και επίσης δεν υπάρχει απαγόρευση αναπαραγωγικού υλικού των ε, κλωνοποιημένων ζώων, δηλαδή σπέρματος και εμβρίων. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της κλωνοποίησης. Τα είπα ήδη, πρόκειται για μια, περι, για μια τεχνική αναπαραγωγής και όχι εκτινοτροφίας, οπότε δεν είναι τροποποίηση γενετική, είναι αναπαραγωγή ενός ζώου που ήδη υφίσταται το πλεονέκτημα είναι πως μπορεί να επιταχύνει την διαδικασία αναπαραγωγής καθώς μειώνεται, μειώνονται ε, οι γενιές, μειώνεται ο χρόνος των γενεών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στους ε, χείρους ε, που υπάρχει ένα σχήμα πυραμίδας και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος χρόνος για να διαχειριστεί ακριβώς το γονίδιο του καλού ζώου. Οπότε έτσι χάνεται ε, ο κίνδυνος να χάσουμε εξαιρετικά πολύτιμα ζώα. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε γονιδιακή ε, επιλογή, όχι τροποποίηση και ήδη έτσι αναγνωρίζουμε την αναπαραγωγική αξία ενός, την κτηνοτροφική με ενός ζώου μόλις έχει γεννηθεί. Μόλις έχει γεννηθεί βεβαίως ε, ένα ζώο όπως ο τάβρος δεν είναι σίγουρο αν θα καταλήξουμε τελικά να έχουμε σπέρμα ή έμβριο από αυτό το ζώο. Εάν λοιπόν ε, διαχυθεί αυτός ο κίνδυνος μέσω της ε, κλωνοποίησης έχουμε πάρα πολλά πλέον εκτήματα στον τομέα της κτηνοτροφίας. Για να συντομεύουμε λοιπόν. για μας είναι αποδεκτή η πρόταση της Κομισιόν, γιατί πρώτα απ' όλα βασίζεται στην αξιολόγηση αντικτύπου της ΕΦΣΑ, σε πολλές αξιολογήσεις αντικτύπου. και βασίζεται σε ε, αρκετά επιχειρήματα υγείας και ευζοίας των ζώων. Βέβαια, δεν έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα, τότε γίνεται με τα ε, έμβρια των κλώνων και καμιά φορά βεβαίως ε, υπάρχουν ζητήματα και στην γέννηση και στο μεγάλωμα των ζώων. Και αισθανόμαστε υπεύθυνοι. Γι' αυτό δεχόμαστε αυτή τη στιγμή την απαγόρευση κλωνοποίηση. Αλλά είναι κάτι το προσωρινό. Γιατί θα πρέπει να αξιολογήσουμε ξανά την κατάσταση σε πέντε χρόνια. Και υποθέτω πως οι επιστήμονες θα λύσουν πολλά από αυτά τα προβλήματα. Και επίση χαιρόμαστε για το ότι δεν απαγορεύεται η έρευνα, η διατήρηση υλικού και των ιατρικών συσκευών. Επιτρέπεται δηλαδή η κλωνοποίηση για αυτά τα ζητήματα αλλά και για την γενετική ποικιλία. Και ξανά το έχω πάλι με κόκκινο δεν απαγορεύεται το αναπαραγωγικό υλικό των ζώων αυτών. Και εδώ πέρα στηρίζουμε την Κομισιόν. Όπως είπα λοιπόν ήδη, Ο περιορισμό αγωγή αναπαραγωγικού υλικού θα είναι κάτι το πολύ κακό για τον κλάδο μας, ε, όχι μόνο για τις εταιρείε αυτές, αλλά και για τους ε, κτηνοτρόφους. Πρώτα απ' όλα θα υπάρχει τεράστιο ε, πρόβλημα, τεράστιο διοικητικό βάρος, θα υπάρχει πρόβλημα ίχνη λασιμότητας, θα υπάρχουν προβλήματα εμπορίου με χώρες όπως η ΕΠΑ, ΕΕ. η συμφωνία TTIP θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά το σημαντικότερο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι το εξή θα επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού σχετικού κλάδου. Θέλω να το τονίσω. Εάν αυτές οι τεχνολογίες και δεν μιλάω μόνο για την κλωνοποίηση. Εάν περιοριστούν αυτές οι τεχνολογίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χάνουμε τη μάχη με τη ΣΥΠΑ. Και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι ε, καινοτόμος, ε, τότε δεν πρέπει να περιορίσουμε αυτές τις εξελίξεις, θεωρώ εγώ. Τώρα, όταν μιλάμε για την πρόταση εμπορίας, ε, η άποψή μας είναι πως η απαγόρευση δεν συμφωνεί με τη γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ. Αυτό είναι σημαντικό ζήτημα για τους κτηνοτρόφους Δεν υπάρχει επίσης περιορισμός ε, προϊόντων απογόνων κλωνοποιημένων ζώων. Και τέλος, όταν η νομοθεσία θα συμπεριλαμβάνει, αν η νομοθεσία αυτή θα συμπεριλαμβάνει και τους απογόνους κλωνοποιημένων ζώων, θα είναι πάρα πολύ αρνητική για τον ε, κτηνοτροφικό τομέα. Τα επιχείρηματά μου είναι τα ίδια με πριν. Η συμβουλή μου λοιπόν είναι πως ίσως δεν είναι ιδανικές οι οδηγίες. Το αντιλαμβάνομαι πως είναι ένας συμβιβασμός. Αλλά για εμάς είναι αυτή τη στιγμή αποδεκτές και θα θέλαμε να συμβουλεύσουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Τουλάχιστον μην τα κάνετε χειρότερα. Μην ενισχύσετε την πρόταση που έφερε η Κομισιόν. Τέλος το όνομά μου εδώ πέρα email, τηλέφωνα, αν θέλετε πληροφορίες είμαι πάντα στην διάθεσή σας. Φένεμαν, παπάκι είμαι στην διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και για την δυνατότητα που μας δίνεται να συνεχίσουμε την συνεργασία και να αξιοποιήσουμε την εμπειρογνωσία σας. Τώρα ο κύριος ε, Ντάβιντ έχει το λόγο, που είναι αντιπρόεδρος της ε, Κόπα Κοζέκα, αρμόδιος για θέματα εκτροφής ζώων. Θα μας παρουσιάσει τη γνώμη της Κόπα Κοζέκα ως προς τις νομοθετικές ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Ξαβία Νταβίτ είναι και διευθυντής του Ινστιτούτου Εκτροφή Ζώων και Τεχνητής Γονιμοποίησης Ζώων στη Γαλλία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας Ε, θα πω δύο λόγια για την κόπα Κοζέκα. Από τη μια πλευρά είναι η κόπα που είναι ε, η Ένωση όλων των ε, συνεταιρισμών ε, ε, γεωργών εκτινοτρόφων και η ΚΟΖΕΚΑ είναι η Ένωση των Ευρωπαϊκών Γεωργικών Συνεταιρισμών. Συμμετέχουν 66 μέλη, οργανώσεις μέλη που αντιπροσωπεύουν περίπου 12 εκατομμύρια γεωργούς και συνεταιρισμούς. Ο στόχος είναι Πρόκειται μάλλον για ε, παραγωγή που ανέρχεται στα 340 δις ετησίως. Ε, στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της γεωργίας και των μελών μας και να βρούμε λύσεις που ε, θα βρίσκουν όλους σύμφωνος. Η πρώτη δήλωση που θα ήθελα να κάνω, το πρώτο πράγμα μάλλον που θα ήθελα να πω, γιατί Έχω ταξιδέψει πολύ στον κόσμο και μπορώ να πω ότι ε, ότι γνωρίζω πως οι Ευρωπαίοι εκτινοτρόφοι σέβονται την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Γίνονται τα πάντα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έχουμε τακτικούς ελέγχους όσον αφορά ας πούμε, την υγεία των ζώων. Έχουμε δις ελέγχου ε, ελέγχους από τις κτηνιατρικές αρχές σε κάθε κράτος μέλο. Δεν συμβαίνει αυτό ε, παντού αλλού. Όσον αφορά την ευημερία των ζώων γνωρίζουμε ότι χωρίς να είναι ε, σε καλή κατάσταση τα ζώα, ποτέ δεν θα έχουμε ε, θετικά τεχνικά ή οικονομικά αποτελέσματα. Ε, αποτελέσματα. Δηλαδή για τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας χρειαζόμαστε τα ζώα μας να είναι σε καλή κατάσταση, να ευημερούν ζωοτεχνική νομοθεσία και πάλι εδώ η νομοθεσία μας γίνεται σεβαστή. συμμετέχουμε στην εκπόνηση κάθε νέας νομοθεσίας και πάλι με στόχο να μπορέσει ε, ο κλάδος μας να παραμείνει ανταγωνιστικός και να μπορέσει να ε, αντιμετωπίσει τη ζήτηση της αγοράς. Το ίδιο και για τα νέα τρόφιμα. Ε, να σας πω επίσης ότι η κλωνοποίηση είναι περιορισμένο ενδιαφέροντος για τους Ευρωπαίους κτηνοτρόφους για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχήν υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά τη γενετική διαφοροποίηση και την ελλειπή γενετική διαδικασία στα ζώα, στα πρόβατα, ε, στις κατσίκες. Δεν χρειαζόμαστε κλωνοποίηση, χρειαζόμαστε αύξηση των διαφόρων ε, ειδών ε, ανάλογα με την μακροβιότητά τους, τη γονιμότητά τους και ούτω καθεξής και Χρειαζόμαστε λοιπόν να έχουμε ε, καλές ράτσες, βιώσιμες ράτσες, αλλά και βιοπικιλότητα. Γι' αυτό και για μας ε, δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεύτερον, δεν γίνεται αποδεκτή η τεχνολογία στην ευρωπαϊκή αγορά. Το αναφέρατε και εσείς στην εισήγησή σας και συμφωνούμε με αυτό. Δεν υπάρχει αποδοχή αυτή τη στιγμή των κλωνοποιημένων ε, ζώων. Δεν θέλουμε τα κλόνους. Ε, δεύτερον, ψηλό κόστος. Μπορείτε να δείτε το Transfora, το website το, ενός μεγάλου αμερικανικού παραγωγού ένα ζώο κοστίζει 20.000 δολάρια. Ε, για να έχεις ένα ζώο, ένα ζώο, ε, νεαρό ζώο ε, κλωνοποιημένο στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται 100.000 ευρώ. Δεν είναι ανταγωνιστική η χρήση του κλώνου, των κλώνων μάλλον, σε, μια, σε ένα αγρόκτημα. Τέλος, χαμηλή αποδοτικότητα. Η έκθεση της ΕΦΣΑ το 2012 έδειχνε αποδοτικότητα μόνο 13 με 25% αν κανείς το συγκρίνει με την γονιμοποίηση in vitro. Μια άλλη άποψη της Κόπα Κοζέκα για την κλωνοποίηση είναι ότι χρειάζεται να συνεχιστεί η έρευνα για τρεις βασικούς λόγους. Για να γνωρίσουμε καλύτερα το μηχανισμό που μας οδηγεί στο να έχουμε καλύτερα και πιο γόνιμα ζώα. Δεύτερον, για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιστημονικών ομάδων στην Ένωση. Και τρίτον, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για μας, είναι ότι η ευρωπαϊκή επιστημονική πυρογνωμοσύνη χρειάζεται ούτως ή άλλως, ειδικά όσον αφορά διεθνή, το διεθνή διάλογο, όπως ας πούμε στο πλαίσιο του ελεύθερου χώρου συναλλαγών υπερατλαντικά, αλλά και γενικά με τρίτες χώρες, εκτός Ευρώπης δηλαδή. Κάτι ακόμα που θέλω να αναφέρω είναι ότι δεν θα πρέπει να υποβαθμίζουμε την κατάσταση, ε, να υποτιμούμε μάλλον την κατάσταση του διεθνού εμπορίου. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι σύμμορφη με όλες αυτές τις νομοθεσίες. Γίνονται διαρκώς ανταλλαγές γενετικών υλικών ανάμεσα στην Ένωση και τρίτες χώρες. Η Ευρώπη δεν είναι νησί, όλοι το γνωρίζουμε. Έχουμε εισαγωγές ε, ε, βοήου κρέατος ή κρέατος, ε, ε, πουλερικών κτλ. Οπότε η πρόκληση για την Ένωση είναι πώς θα συμφιλιώσει τρεις, τρία βασικά ζητήματα. Πρώτον, δίκαιος ανταγωνισμός ανάμεσα στην βιομηχανία ε, κτηνοτροφίας στην Ένωση, πώς ε, θα υπάρξει κοινωνική αποδοχή που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τους ευρωβουλευτές αλλά και πώς θα γίνει, θα εξασφαλιστεί η ε, ανιχνευσιμότητα. Τέλος, η Κόπα Κοζέκα θα προτιμούσε ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Ε, τώρα, ποιο νομικό μέσο είναι το καταλληλότερο, οδηγία ή κανονισμός. Εμείς πιστεύουμε ότι κανονισμός είναι καλύτερος γιατί μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα για όλες τις χώρες ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου. Ε, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει ανιχνευσιμότητα για τους κλόνους που κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Αλλά για τους απογόνους των κλόνων πολύ πιο δύσκολο θα είναι, γιατί θα χρειαστεί μια κεντρική βάση δεδομένων που είναι πολύ δαπανηρή και περίπλοκη και σύμφωνα με την έκθεση της ΕΦΣΑ δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους κλόνους και τους απογόνους τους. Κάτι ακόμα ε, είναι ότι η ανιχνευσιμότητα στα μεγάλα ζώα είναι πολύ δαπανηρή. Ε, έγινε κάποια συζήτηση σε σχέση με την ανιχνευσιμότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ηλεκτρονικό, την ηλεκτρονική ταυτότητα και η Επιτροπή, η Ευρώπη είπε να μην το καταστήσει αυτό υποχρεωτικό στα μεγάλα ζώα, ακόμα και αν ε, είναι ενδιαφέρουσα ε, η θέση και αυτό μόνο και μόνο λόγω του κόστους. Η, ε, η ατομική ηλεκτρονική ταυτότητα είναι πολύ δαπανερή και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην Ευρώπη. Τελευταία παρατήρηση για την κόπα Κοζέκα που θέλω να αναφέρω πιο λεπτομερώς είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει διάκριση κατά εμάς ανάμεσα στους κλόνους και τους απογόνους τους και γι' αυτό και θέτουμε επιτάπητος και πάλι την γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ ως προς αυτό το θέμα είναι σαφέστατη. Τώρα όσον αφορά την διαφοροποίηση ότι οι απόγονοι δεν έχουν διαφορές με τους συμβατικούς απογόνους για μας αυτό δεν ισχύει και η κλωνοποίηση δεν είναι θέμα μόνο ασφάλειας τροφίμων. Τέλος, ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να εγγυάται την απουσία κλώνων ή απογόνων αυτών στη ζώα του. Πώς θα το κάνει αυτό αν δεν έχει τις απαραίτητες πληροφορίες, εάν η τρίτη, το τρίτα μέρη δεν είναι διαφανή και ποιος θα πληρώσει για την ανάπτυξη ακατάλληλων μεθόδων ελέγχου, ποιος θα επομιστεί το κόστος Γι' αυτό συμφωνούμε με την πρόταση της Κομισιόν σε αυτή τη φάση, ότι δηλαδή δεν έχουμε εμείς καμία ιδιαίτερη χρήση για τους κλόνους από την πλευρά των Ευρωπαϊκών Κοινοτροφικών Εταιριών για στόχους διατροφής, κατασκευής τροφίμων. Μάλιστα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ντόναλτ Μπρουμ, που είναι επίτιμος καθηγητής για την ευημερία των ζώων στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Μάλιστα, ο κύριος Μπρούμ έχει επεξεργαστεί πολλές επιστημονικές μεθόδους για τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Δημοσίευσε πάνω από 300 άρθρα για θέματα ευημερίας των ζώων και εργάστηκε σε πολλές επιτροπές σχετικές της Μεγάλης Βρετανίας και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μάλιστα ήταν για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευημερία των Ζών και μέλος του επιστημονικού πάνελ της ΕΦΣΑ. Είναι και πρόεδρος της Ειδικής Ομάδας για την Ευημερία των Ζών κατά τη μεταφορά τους. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς ο κύριος Μπρουμ. Όπως ακούσατε είμαι επιστήμονας αρμόδιος, ειδικός ε, για την ευημερία των ζώων. Δεν εκπροσωπώ καν μία οργάνωση, δεν είμαι μέλος καμίας οργάνωσης προστασίας των ζώων ή χρήστης ε, εκτροφέας. Ε, ήμουν πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ε, για, για την Ευημερία των Ζώων μεταξύ του 1990 και του 2009 και μέλος του Πάρελ της ΕΦΣΑ. Το, η ευημερία των ζώων είναι μια κατάσταση που αφορά την προσπάθεια του ζώου να αντιμετωπίσει το περιβάλλον του. Και ποικίλει από, τι πολύ κακή, από τις πολύ κακές συνθήκες διαβίωσης και μπορεί να εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί επιστημονικά. Το θέμα είναι πώς λειτουργεί το ζώο ε, στο περιβάλλον του και αν είναι σωστό να αλλοιώνουμε τις φυσικές διαδικασίες. Ο κλωνοποίηση των ζώων γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Τα πρώτα ζώα κλωνοποιήθηκαν το 1950, τα αμφίβια, ενώ τα θηλαστικά κλωνοποιήθηκαν το 1986 όπως θα γνωρίζετε μάλλον, άλλο κλωνοποίηση και άλλο γενετική μετάλλαξη. Γιατί η γενετική μετάλλαξη προϋποθέτει νέο γενετικό υλικό, ενώ η κλωνοποίηση δεν ε, προσθέτει νέο γενετικό υλικό στο, γονό, στο γονιδίωμα. Η βασική διαδικασία που χρησιμοποιείται είναι το SCNT, δηλαδή πυρηνική μεταφορά σωματικού κυτάρου. Αυτή είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται κατά εξοχήν για την κλωνοποίηση. Τα αποτελέσματα των διαδικασιών κλωνοποίησης ε, είναι πολλά και διάφορα. Μερικά είναι αρνητικά και άλλα θετικά. Τα αρνητικά στην ε, ευημερία των ζώων αφορούν τη μητέρα. Υπάρχουν όμως κάποιες παρενέργειες που αφορούν τον απόγνο, το ζώο. Ε, κυρίως όταν το κύτταρα αναπτύσσονται σε ένα ε, ζώο όταν είναι νεαρό και όταν ενηλικιώνεται και επίσης επηρεάζει και τους απογόνους, τις ε, μεταγενέστερες, επερχόμενες γενναίες ε, που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα ε, είτε ένα αμετάβλητο περιβάλλον είτε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Επίσης κάποια αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία τους ή και σε άλλα ζώα που δεν έχουν κλωνοποιηθεί. Ε, βέβαια με την κλωνοποίηση μειώνεται ο αριθμός των ζώων που χρειάζονται για αναπαραγωγή. Τώρα η απόχωνη των κλωνοποιημένων ζώων, μάλιστα όταν κλωνοποιείται ένα ζώο και έχει περάσει το νεαρό στάδιο, το περισσότερα ζώα κανονικά αντιμετωπίζουν το περιβάλλον τους επιτυχημένα, παρόλο που έχουν εντοπιστεί κάποια προβλήματα. Οι επερχόμενες γενές προς το παρόν δεν ξέρουμε πώς αντιμετωπίζουν ε, το περιβάλλον και αν επηρεάζονται αρνητικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα. Απλώς δεν έχουμε αποδείξεις για κάτι τέτοιο. Γίνονται μελέτες αλλά δεν έχουμε τεκμήρια. Πάντως, αν τα ζώα κλωνοποιείται είναι υψηλή παραγωγικότητα, τέτοια ζώα ε, διαβιούν σε χειρότερε συνθήκε από ότι τα ζώα που έχουν χαμηλή παραγωγικότητα. Και άρα αυτό επηρεάζει την ευημερία του κυρίω στι επερχόμενε γενιέ. Αντίθετα δηλαδή με τα άρθρα 20 και 21 τη οδηγια 98 98-58. Οπότε ε, ταχαίως αναπτυσσόμενα κοτόπουλα για κρεατοπαραγωγή διαβιούσε χειρότερες συνθήκες ε, με ασκήτη, ε, παθήσεις ε, στα πόδια, εγκάβματα στον ταρσό, φλίκτενες στο στήθος, ενώ αγελάδες κλωνοποιημένες μπορούν να παρουσιάσουν μαστίτιδα, παθήσεις στα ζώα και αναπαραγωγικές διαταραχές. Παθήσεις στα πόδια και Αναπαραγωγικέ διαταραχέ. Τώρα, αν δούμε πώς προσπαθούν τα ζώα να αντιμετωπίσουν το περιβάλλον τους, βλέπουμε ότι αν περιορίζουμε τη γενετική πολυμορφία, θα δυσχεράνουμε την προσαρμοστικότητα των ζώων στις νέες συνθήκες. Για παράδειγμα, αν εμφανιστεί μια νέα νόσος, μια νέα επιζωτία, η γενετική ομοιομορφία αυξάνει τον κίνδυνο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης μιας νέας νόσου. Οπότε δεν χρειαζόμαστε πολύ γενετική ομοιομορφία. Γιατί κάτι τέτοιο αποδυναμώνει τα ζώα και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν οι Ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι. Πολύ συχνά είχαμε νέε επιζώτιες τα τελευταία χρόνια. Κάτι που ίσως δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον, γιατί το περιβάλλον αλλάζει, η θερμοκρασία, έχουμε τις κλιματικές αλλαγές. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα κλωνοποιημένα ζώα. Επίση, αν έχουμε εξάπλωση μια νέα επιζωοτία εξαιτία τη μειωμένη προσαρμοστικότητα των ζώων, αυτό θα επηρεάσει το σύνολο των ζώων. Όχι μόνο τα κλωνοποιημένα ή του απόγονου κλωνοποιημένων. Του απογόνου, συγγνώμη, κλωνοποιημένων. Τώρα, υπάρχουν κάποιε θετικέ ε, συνέπειε από την κλωνοποίηση. Ξέρουμε ότι τα ζώα που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή ίσως διαβίωσε σε χειρότερες συνθήκες, γιατί κυρίως είναι από ράτσα που αναπτύσσεται γρήγορα και άρα ε, υποβάλλονται σε επισητιστικούς περιορισμούς για να μην μεγαλώνουν τόσο γρήγορα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βέβαια, έτσι με την κλωνοποίηση μειώνουμε τα προβλήματα και από αυτή την άποψη μειώνοντα τα ζώα αναπαραγωγής που χρειαζόμαστε θα έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα, όχι όμω άμεσα. Γιατί η αποτελεσματικότητα τη κλωνοποίηση προ το παρόν είναι πολύ χαμηλή. Οπότε μπορεί να είναι κάτι πιθανό για το μέλλον, αλλά δεν είναι ακόμη δυνατό σήμερα. Τώρα για όλα τα θηλαστικά και τώρα περνώ στα άμεσα αποτελέσματα στις μητέρες και τα ζώα που γεννιούνται, που είναι κλωνοποιημένα, ενώ όταν γίνεται πυρηνική μεταφορά σωματικού κυτάρου, δημιουργείται ένα έμβριο που ε, μεταφέρεται σε παρένθετο ζώο και αυτό, όταν το έμβριο επιβιώνει δεν ε, έχει αρνητικές συνέπειες στις συνθήκες διαβίωσης. Το πρόβλημα για τη μητέρα και για το νέο ζώο ή το νέο ζώο που κλωνοποιείται είναι ότι αυτή η πυρηνική μεταφορά σωματικού κυτάρου δημιουργεί ανομαλίες του πλακούντα και πολλές φορές και ανομαλίες ή ε, δυσμορφίες του εμβρίου. Μπορούμε να έχουμε ένα υπερβολικά μεγάλο έμβριο στην μητέρα ή να δημιουργηθούν διαταραχές στον πλασέντα και να μην μπορέσει ε, το ζώο να γεννήσει. Κάτι που είναι αρνητικό ε, για το ζώο που γεννά. Και επίσης αν έχουμε δυσμορφία του εμβρίου ε, θα έχουμε αρνητικά αποτελέσματα για το ζώο που θα γεννηθεί. Οπότε όλα αυτά είναι αρνητικά για την ευημερία του ζώου. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για όλα τα ζώα, αλλά για μεγάλο ε, τμήμα των ζώων, κάτι που δεν θα είχαμε με κανονικές μεθόδους εκτροφής και αναπαραγωγής. Τώρα, μπορούμε με νέες τεχνολογίες να βελτιώσουμε τη διαδικασία αυτή. Μία άλλη πρόταση γίνεται από μια ομάδα στην Ιαπωνία, τους Βατανάμπη και Ναγκάι, που δήλωσαν ότι δεν έχει βελτιωθεί η συχνότητα των βλαβών ε, μεταξύ 1998 και 2007. Ούτε και από το 2007 όμως έχουμε βελτίωση. Εδώ και πολύ καιρό η τεχνολογία είναι προβληματική και δεν έχει βρεθεί άλλη καλύτερη μέθοδος από την πυρηνική μεταφορά σωματικού κιτάρου. Υπάρχουν όμως και άλλες μέθοδοι, αλλά στο, προς το παρόν δεν κρίθηκαν καλύτερες από τις υπάρχουσες ή από τις προϋπάρχουσες. Τώρα, για τα μεμονωμένα είδη, για τα, βο, τα, οι κλόνοι βοηδών έχουν υψηλό βαθμό θνησιμότητας πολλά έμβρια πεθαίνουν σε πολύ πρώιμο στάδιο ή μετά τη ε, διαμόρφωση του ε, εμβρίου, 27% μόνο των, ε, των ε, εγγύων ζώων καταφέρουν να γεννήσουν και μάλιστα ακόμη χειρότερη κατάσταση είναι για το υδροβούβαλο. Κάτι που δεν έχουμε σε κανονικές μεθόδους αναπαραγωγής έχουμε πολλές δυσμορφίες εξαιτία της κλωνοποίησης και παθολογίες που διαπιστώσαμε σε κλωνοποιημένα ζώα. Έχουμε σημαντικές λοιπόν συνέπειες αρνητικές και με τη μητέρα και για το ζώο που γεννιέται. Μετά την νεαρή ηλικία μειώνονται τα προβλήματα, αλλά έχουμε μείωση της διάρκειας ζωής. Ε, τα γουρούνια και τα εγωπρόβατα χρειάζονται χειρουργική επέμβαση για να γίνει η μεταφορά του πυρήνα από το ο κύτταρο. Πολύ πιο παρεμβατική διαδικασία, κάτι που επηρεάζει την ευημερία. Επίσης έχουμε αύξηση της θνησιμότητας των εμβρίων στους χείρους και μειωμένη διάρκεια ζωής στους χείρους. Αλλά δεν είχαμε μεγάλο δείγμα. Για τα πρόβατα έχουμε δυσμορφίες αντίστοιχες με αυτές που έχουμε και στα βοηδή. Σημαντική μείωση του αριθμού των αγγεία της εγκυμοσύνης και λίγα είναι τα πρόβατα που επιζούν μετά τον απογαλακτισμό. Τώρα για τα πτηνά. Προς το παρόν δεν έχει επιτευχθεί πλήρης κλωνοποίηση. Όταν γίνεται όμως ε, μεταφορά των ε, αρχαίων μεταμόσχευση μάλλον των αρχαίων γεννητικών κυτάρων, έχουμε κάποια στοιχεία. Είχαμε τρεις ε, μελέτες με ποσοστό εκόλεψη όμως μόνο 3% επιβίωση και 77% μετά την γέννηση. Σημαντικά αποτελέσματα στα πτηνά. Τώρα στα ψάρια έχουμε τα ίδια προβλήματα. Και στα ψάρια η χθιοτροφή το πρόβλημα είναι μείζον ζήτημα, αλλά δεν αντιμετωπίζεται από το πρώτο έγγραφο, την πρώτη πρόταση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κλωνοποίηση των ψαριών οδηγεί σε προβληματικά ε, ψάρια με πολλές δυσμορφίες. Οπότε η κλωνοποίηση στα ψάρια είναι και ιδιαίτερα προβληματική. Ποια είναι τα συμπεράσματα τώρα, τα επιστημονικά πορίσματα για την ε, ευημερία στις, ε, στα ζώα μητέρες και στους απογόνους είναι αρνητικά. Ε, για τα θηλαστικά, τα πτηνά και τα ψάρια. Δεν υπάρχει εναλλακτική προς το παρόν ε, μεθοδολογία να αντικαταστήσει τις τρέχουσες διαδικασίες και δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι στο μέλλον θα εφευρεθούν νέες μεθοδολογίες. Οπότε η αύξηση της γενετικής ομοιομορφίας θα έχει αρνητικές συνέπειες στην προσαρμοστικότητα των ζώων σε νέες ασθένειες. Επίσης, ό,τι αφορά την ευημερία των ζώων έχουμε πολύ περισσότερα αρνητικά από ό,τι θετικά αποτελέσματα και αυτό και ο γενικός απολογισμός είναι αρνητικός. Τώρα, το γεγονό ότι τρόφιμα από ζώα δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι επιζήμια για την ανθρώπινη υγεία, ε, το κοινό είναι αρνητικό εξαιτία ε, ε, των αρνητικών συνεπειών στην ευημερία των ζώων. Για σκεφτείτε χείρι που ε, είναι σταυλισμένοι και δεμένοι σε πολύ αρνητικέ συνθήκε. Ο κόσμο δεν θέλει να καταναλώσει τέτοιο χείρινο κρέα, γιατί ξέρουν ότι το ζώο έχει ταλαιπωρηθεί. Όπως ο κόσμος δεν αγοράζει προϊόντα με δέρμα φώκες επειδή ξέρουν ότι έχουν βασανιστεί οι φτώχε για να γίνει εκδορά του, Όχι επειδή τα προϊόντα από δέρμα φώκιας κατά ανάγκη είναι επιζήμια για την υγεία. Οπότε ο κόσμος αποφύγει να αγοράσει ε, γενιές ε, ή απογόνους κλωνοποιημένων ζώων και θα έχει ιδιαίτερε απαιτήσει για την ετικετοθεσία τέτοιων προϊόντων. Το 2013 ε, είχαμε τον κανονισμό 0433 για τα τηλαστικά και το, τον κανονισμό 0434 που αφορά γενικώ τα ζώα και άρα θα περιλάμβανε και τα ψάρια. Επειδή είναι παρόμοιε οι επιστημονικέ αποδείξει ε, για τι κακέ συνθήκε διαβίωση ε, θηλαστικών ψαριών και ε, πτηνών, πιο λογικό θα ήταν να έχουμε όλα τα ζώα στην ίδια κατηγορία και δεν βλέπω το λόγο να υπάρχει διαφοροποίηση των δύο κανονισμών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Μας δώσατε μια επιστημονική σκοπιά και σκοπιά, τη σκοπιά της φυσιολογίας έχουμε εμπλουτίσει τις γνώσεις μας και με πολύ σημαντικές επιστημονικές πληροφορίες. Και θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γιλέρα. Παρακαλώ. 1,5 λεπτό καθένας παρακαλώ. Περιοριστείτε σε ερωτήσεις προς τους επιφανείς εμπειρογνώμονές μας. Κυρία Γιλέρα, παρακαλώ 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι και σκιώδη συγγήτρια της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Γι' αυτό και παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, την δημόσια αυτή ακρόαση που περίμενα και με αδημονία, γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι σημαίνει κλωνοποίηση και ποιες είναι οι συνέπειές της. Δεν το γνωρίζουν ούτε οι πολίτες, αλλά ακόμη και εμείς. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε τα επιμέρους ε, στοιχεία αυτού του περίπλοκου θέματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις εμπειρογνώμονές μας για τις παρουσιάσεις τους που κατέληγαν σε διαφορετικά ίσως συμπεράσματα αλλά ήταν όλες ενδιαφέρουσες. Όπως είπε και ο Πρόεδρος θα πρέπει να περιοριστούμε σε ερωτήσεις. Ερωτώ λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σας για το άρθρο 3 των δύο προτάσεων. Γιατί το άρθρο 3 αφήνει στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών να εξασφαλίσουν τη μη εισαγωγή στην αγορά τους παράγων προϊόντων από κλωνοποιημένα ζώα. Δηλαδή το κράτος μέλος θα πρέπει να οριοθετεί κατά κάποιο τρόπο τα σύνορά του. Κατά τη γνώμη σας, και κατά τη γνώμη του καθηγητού, του επιστήμονα, πιστεύετε ότι είναι δυνατό τα κράτη-μέλη να προβλέψουν διαφορές και να οριθετήσουν τα σύνορά τους. Είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Το θεωρείτε εφικτό. Ευχαριστώ. Κύριος Φεράντ. Φεράντ. Φερό, συγγνώμη. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το περασμένο Δεκέμβριο είχα ήδη παρέμβει για αυτό το θέμα όσον αφορά την νομοθεσία για την κλωνοποίηση που είχε παρουσιαστεί εδώ ε, σε αυτή την Επιτροπή και είχα υπογραμμίσει κάποια προβλήματα. Καταρχήν ε, τον αποκλείονται ε, οι απόγονοι αλλά και οι η ταξινόμηση των συναλλαγών με χώρες που κάνουν κλωνοποίηση, αλλά και αδυναμία πραγματικού και αξιόπιστου ελέγχου ε, στις εισαγωγές. Έχω λοιπόν να, εκφράσω κάποιες, να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Γιατί να επιμένουμε να συζητάμε για ένα θέμα που είμαστε σύμφωνοι εδώ στην Επιτροπή Άγκρη. Δυστυχώς πιστεύω πως γνωρίζω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα πρέπει και πάλι, μάλλον ακόμα μια φορά η όθηση για η βούληση για να προωθηθούν νομοθεσίες ε, συμβατές με αυτές των Ηνωμένων ε, Πολιτειών που αυτές ε, έχουν, κάνουν χρήση της κλωνοποίηση. Εμεί, μήπω εντάσσεται μάλλον αυτή η συζήτηση στην προετοιμασία των διαπραγματεύσεων για την TTIP. Και αυτό δεν θυμίζει το ατυχές προηγούμενο των γενετικά τροπομένων οργανισμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μηχανή που σέβεται τα αιτήματα των πολιτών της, των λαών της και των ε, κλεγμένων της εκπροσώπων. Είμαστε το τελευταίο αστεράκι της Αμερικανικής σημαίας. Και να θυμίσω στον κύριο ε, Νταβίντ ε, που ότι ως Γάλλος προτιμώ να είχε πάρει το λόγο στη γλώσσα του Μολιέρου, αφού είναι Γάλλος. Ευχαριστώ. Παρακαλώ ερωτήσεις να υποβάλλετε προς τους εμπειρογνώμονές μας. Ο κύριος Λαζού. Pan Λαζού. Oui, nous sommes évidemment... Euh, Είμαστε παντελώ αντίθετοι στην κλωνοποίηση ζώων κτηνοτροφία, διότι η γενετική χειραγώγηση και η κλωνοποίηση δημιουργούν προβλήματα για τα ίδια τα ζώα που έχουν κλωνοποιηθούν ή γενετικά τροποποιηθεί, ιδιαίτερα για τι μητέρε που τα φέρουν μέχρι τη γέννησή του με ποσοστά σε πολύ ψηλά, καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα. Στη θεωρία αυτές οι τεχνικές δεν είναι φυσιολογικές και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία των ζώων. Συνέπεια καταρχήν είναι ε, να γίνονται δύσκολες οι, ε, οι δύσκολοι τοκετοί, ε, αυξημένη ευαισθησία στις μεταδοτικές ασθένειες, 10% περίπου γεννιέται και ανάμεσα σε αυτούς, αυτά από τα ζώα που γεννιούνται, κάποιοι πολλά δεν επιβιώνουν στον απαγαλακτισμό. Δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικές, δε οι τιμές. Άρα λοιπόν ρωτώ, Πρόεδρε, και εσάς τους με βάση όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν, δεν θα έπρεπε πια να σκεφτούμε να εγκαταλείψουμε αυτή την πολιτική τρέλα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γλέζος. Αγαπητοί πρόεδροι, συμπρόεδροι, αγαπητοί συγητές και συνάδελφοι. Νομίζω ότι το θέμα εξετάστηκε με εξαιρετικές μονάχα περιπτώσεις μονάχα από την οικονομική του πλευρά, από την οικονομική του διάσταση. Δηλαδή αν συμφέρει στον άνθρωπο, αν είναι ανταγωνίσιμο, εάν τα προϊόντα που δημιουργούνται μπορούμε ή δεν πρέπει να τα τρώμε. Και δεν εξετάστηκε στη βασική του θεμελιακή αντίληψη των σχέσεων του ανθρώπου μας με τη φύση. Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε πάνω από τη φύση ούτε έξω από τη φύση, ούτε κάτω από τη φύση. Είναι δημιούργημα της φύσης. Και ως δημιούργημα της φύσης ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτιάξει φυσικούς νόμους, μπορεί να αξιοποιήσει τους φυσικούς νόμους. Εάν δεν δούμε όλη αυτή την τοποθέτηση θα πελαγοδρομούμε στα συμφέροντα εάν το προϊόν μπορούμε να το φάμε ή όχι, εάν είναι ανταγωνίσιμο ή όχι. Γι' αυτό το λόγο, με την κλωνοποίηση, τι προσπαθούμε να κάνουμε, να διορθώσουμε τη φύση, για σκεφτείτε το αυτό. Και επειδή τελευταία στην Ελλάδα έγιναν εκλογές και τώρα στο Eurogroup συζητιέται πάρα πολύ το θέμα της Ελλάδας διαβλέπω μια καινούργια προσπάθεια κλωνοποίησης της Ελλάδας. Όχι την Ελλάδα όπως τη γνωρίζετε και τι θέλετε να είναι, αλλά προσπαθούν οι δανειστές της να την κλωνοποιήσουν. Την εμποδίζουν να αποκτήσει την εθνική της ανεξαρτησία, την εμποδίζουν να βγάλει τη θηλιά από το λαιμό που τις έχουν φορέσει οι δανειστές της. Εμποδιστε την κλωνοποίηση της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ. Πολύ εύστοχα το θέσατε. Κυρία Μιλερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτά τα οποία είπατε και είπαν και οι ειδικοί. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα. Θα ήθελα να μας πει ο Επίτροπος ε, πότε θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της μελέτης. Εγώ θα ήθελα να τα λάβουμε σύντομα και μετά ποια είναι ε, η οικονομική σημασία των εξαγωγών τρίτων χωρών προς την Ένωση για αναπαραγωγικό υλικό, για σπέρμα, τι επιπτώσεις έχει αυτό εάν ε, όντως ε, απαγορεύσουμε κάτι τέτοιο. Και άλλο ένα ερώτημα προς τον κύριο Φένεμαν. Μιλήσατε για το TTIP και το τι θα μπορούσε να σημάνει αυτό. Έχετε επίσης κάποιες επιφυλάξεις ε, ε, για την γενετική ποικιλία. Εγώ είμαι κτηνοτρόφος και δεν θέλω την κλωνοποίηση για λόγους ε, ηθικούς, όχι για κάποιον. Ο κύριος ähm, ich Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό το οποίο υπόθηκε. Πρόκειται για μια τεχνολογία περιττή, την οποία δεν θέλουμε στην Ευρώπη. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Για το ποσοστό των δυσμορφιών ε, στην ε, διαδικασία αυτή. Εγώ θεωρώ πως θα πρέπει να απαγορεύσουν αυτή τη διαδικασία χωρίς ε, καμία συζήτηση για αυτό τον ε, λόγο και μόνο. Και νομίζω πως αν μας δώσετε και τα ποσοστά των δυσμορφιών θα έχουμε άλλον έναν λόγο. Αλλά κάτι άλλο προς την ε, Κομισιόν. Όταν μιλάμε για εισαγωγές ε, δεύτερης γενιάς κλώνων, γιατί μας λέτε πως θα πρέπει να γίνει αυτό για λόγους ε, κόστους, αλλά δεν έχετε υπολογίσει το κόστος. Και μας λέτε θα φέρουμε μία μελέτη. Μα τέσσερα χρόνια το συζητάμε. Πού είναι αυτή η μελέτη. Η υποψία μου και το είπε νομίζω και ο πρώτος ομιλητής είναι πως θέλετε απλά να αποφύγετε τις συγκρούσεις με τις ΗΠΑ λόγω της ε, συμφωνίας ε, της Διατλαντικής. και μετά μας λέτε πως θα είναι μεγάλο το, το κόστος. Κοιτάξτε, είναι απλό. Αν εμείς αποφασίσουμε πως δεν θέλουμε την κλωνοποίηση, το ίδιο ισχύει και για τους απογόνους των ε, κλώνων. Οπότε δεν είναι συνεπής εδώ πέρα η άποψη της ε, Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε σε αυτή την θέση ως ε, Κοινοβούλιο, θεωρώ εγώ. Ευχαριστώ κύριος Μποβέ. Ευχαριστώ. Καταρχήν θερμά ευχαριστώ στους εμπειρογνώμονες ε, για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που μας έκαναν. Νομίζω ότι το πρώτο ερώτημα που ανακύπτει είναι αν σήμερα χρειαζόμαστε πραγματικά ζώα που έχουν αναπαραχθεί ε, με κλωνοποίηση. Αν αυτό είναι προς το συμφέρον της εκτινοτροφίας. Αυτό πρέπει να δούμε πρώτα, το συμφέρον μας. Έχουμε μια πολυμορφία στην παραγωγή. Δεν χρειαζόμαστε κλόνους σήμερα. Ερωτώ λοιπόν, προς τι οι κλόνοι τους χρειαζόμαστε. Γιατί αν δεν του χρειαζόμαστε, γιατί κλωνοποιούμε τα ζώα. Ποιον εξυπηρετεί η κλωνοποίηση. Πολλοί μίλησαν για τις ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Θα ήθελα στην έκθεσή μας και στην ε, απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα πούμε καθαρά και εξάστερα. Δεν θέλουμε ε, εισαγωγές από χώρες που επιτρέπουν κλωνοποίηση αν δεν έχουμε το DNA των κλωνοποιημένων ζώων, των, ε, ζώων, των μητέρων ζώων και των απαγόνων, Θα πρέπει να ελέγχουμε όλα τα ζώα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγουμε την εισαγωγή κλωνοποιημένων ζώων. Γιατί σήμερα λέμε εύκολα ετικετοθεσία. Πώς θα κάνουμε την ετικετοθεσία. Πρέπει να έχουμε ένα ένα μικροτσίπ για να γνωρίζουμε ποιο είναι το DNA του αρχικού ζώου και του απογόνου. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Επίσης, μιλήσαμε για επιζωτίες, μιλήσαμε για δυσμορφίες ε, ή παραμορφώσεις. Θα ήθελα ο επιστήμονας να μου με ρωτήσει. κάνουμε πολλούς ε, πολλαπλασιασμούς ε, του υλικού για να έχουμε, να καταλήξουμε στο καλό κλόνο, που σημαίνει εντατικές ορμονικές θεραπείες προς τις μητέρες, κάτι που δημιουργεί άλλο πρόβλημα υγείας, γιατί έχουμε αποδυνάμωση και φοβερή κακοποίηση του ζώου. Ας μην το ξεχνούμε και αυτό. Και τέλος, γιατί δεν ξέρω αν έγιναν αναλύσεις σχετικά, τα, τα προϊόντα των ζώων, το γάλα για παράδειγμα, ε, παρουσιάζει διαφορές στο μεταβολισμό του ανάλογα με το αν προέρχεται από κλωνοποιημένο ζώο ή όχι. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Χάζακαμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σοκάρομαι ότι ε, πάλι συζητάμε για την κλωνοποίηση. Οι καταναλωτές δεν τη θένε, οι κτηνοτρόφοι δεν τη χρειάζονται και τα ζώα υποφέρουν πάρα πολύ. δεν είναι μόνο ακριβή και χρειάζονται και πάρα πολλά ζώα ούτως ή άλλως για να εφαρμοστεί. Χρειαζόμαστε κάποιες παρένθετες μητέρες, κάποιες μητέρες θα δώσουν το γενετικό υλικό και πάρα πολλά πράγματα. Ε, αυτό είναι το σκεπτικό, αλλά άμα δει κανείς την ιστορία αυτή και το ερώτημά μου επευθύνεται προς τον δόκτωρα Μπρούμ. Βλέπετε πως ε, αυτή η υπόθεση έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιες δεκαετίες. Και πραγματικά στην παρουσίαση αυτή δεν κατάλαβα εάν έχει υπάρξει κάποια βελτίωση στην τεχνολογία, στη μεταχείριση των ζώων, και παρόλα αυτά άκουσα κάποιες βουλευτές να ζητάνε ένα προσωρινό μονατόριο μου αντί για πλήρη απαγόρευση. Ερωτώ λοιπόν, θεωρείτε πως θα υπάρξει κάποια βελτίωση της ε, τεχνολογίας ε, στο προσ... Ευχαριστώ. Dziękuję pan Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Μπέλντερ. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Πρώτα απ' όλα να πω πως ε, το κόμμα μου ε, ως χριστιανικό κόμμα είναι κατά της ε, κλωνοποίησης για ηθικούς λόγους. και κατόπιν ε, το συγκεκριμένο ερώτημα προς τον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν. Αναφέρω από την πρότασή σας. Λέει, διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων είπα και Αργεντινή είπαν πως στο εδαφός τους κλωνοποιούνται ζώα, αλλά δεν μπορούσαν να μας πούν σε ποιο βαθμό συμβαίνει αυτό. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Είναι ανησυχητικό οι εμπορικοί μας εταίροι να μην μπορούν να δώσουν μια απάντηση όταν η κλωνοποίηση έχει τόσο σοβαρές συνέπειες. Αναμένω λοιπόν μια απάντηση από την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Αγίουζο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονές μας. Αντιλαμβάνομαι ότι η κλωνοποίηση βελτιώνει τη γενετική και είναι κάτι που μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και η επιστήμη και ότι δεν δημιουργεί η κλωνοποίηση κανένα πρόβλημα για την επιστημιστική ασφάλεια. Σε λίγο θα ακούσουμε και την ΕΦΣΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων. Περισσότερο τα προβλήματα είναι ηθικά, διοντολογικά και θέματα ευημερίας των ζώων ή καλής διαβίωση των ζώων. Αυτό που με ανησυχεί είναι μία, ε, μία πρόταση ε, ετικετοθεσίας. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να, κάνουμε, να βάζουμε ετικέτες ε, στα κλωνοποιημένα ζώα, αλλά πώς θα κάνουμε τη διαφοροποίηση μεταξύ των απογόνων. Γιατί είναι σαν δίδυμα ουσιαστικά αυτά τα ζώα. Πώς θα κάνουμε την ετικετοθεσία στις επερχόμενες γενναίες. Γιατί μια τέτοια προσπάθεια δικαιοθεσίας και θα είναι και σχεδόν ανέφικτη. Επίσης, πώς θα αποφύγουμε εισαγωγή σπέρματος κλωνοποιημένων ζώων. Γιατί είναι εύκολο κανείς να το φέρει και σε ένα σωλήνα ακόμη και στη βαλίτσα του. Euh, Ο κύριος Αντρίε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Επίτροπο και τους εμπειρογνώμονες. δεν θα πρωτοτυπήσω σε σχέση με τους προλαλήσαντες. Σήμερα στην ακρόαση ακούσαμε τρεις εμπειρογνώμονες και δεν ακούσαμε πιστικά τουλάχιστον επιχειρήματα που να δικαιολογούν αναπαραγωγή ζώων με κλωνοποίηση. Μιλήσαμε για αναπαραγωγικό υλικό, σπέρμα και έμβρια και απογόνους δεύτερης γενιάς. Αυτά τα στοιχεία είναι προβληματικά, το ακούσαμε. Και η κλωνοποίηση δημιουργεί προβλήματα. Μας τα είπε ο επιστήμονας. Προβλήματα στην ευημερία των ζώων. Τώρα, ούτε η ετικετοθεσία είναι επαρκής λύση. Και μερικές φορές και ανέφικτη. Ερωτώ λοιπόν, τι δικαιολογεί σήμερα. Ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την συνέχιση των ερευνητικών εργασιών, των ερευνών για την κλωνοποίηση. Μετά από όλα αυτά που ακούσαμε, ακούσαμε και από τους ευρωβουλευτές, αλλά και από τους επιρρογνώμονες. Γιατί ακούσαμε κάποιους ε, υπενιγμούς για διαδικασίες ε, ή για νομολόγητους στόχους ε, σε ό,τι αφορά τη συνέχιση των εργασιών για την κλωνοποίηση. Σίγουρα η επιστήμη θα μας τα πει αυτά. Η κυρία Σένερα. Η κυρία Σένερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες, τους καλεσμένους μας. Και μετά από πολύ προσεκτική ακρόαση των παρεμβάσεων, θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό επιβεβαιώνεται κάτι που γνωρίζαμε ήδη. Ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε με την κλωνοποίηση. Προς τι η κλωνοποίηση. Έτσι, μόνο αυξάνουμε το κόστος παραγωγής των κτηνοτρόφων. Εκτός αν υπάρχει και κάτι που υποβόσκει, κάτι ανομολόγητο. Αλλιώς γιατί να χάνουμε χρόνο και χρήμα σε συζητήσεις για κάτι που όλο και πιο σαφώς προκύπτει ότι είναι άχρηστο και ακατάλληλο για την κοινωνία και για τους πολίτες. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από την προσπάθεια συνέχισης και προώθησης του ζητήματος κλωνοποίησης. Ευχαριστώ. Κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, όταν άκουγα τους διάφορους εμπειρογνώμονες που παρενέβησαν προηγουμένως και τους οποίους ευχαριστώ, σκέφτηκα, μα γιατί γίνεται αυτή η ακρόαση αφού Ακόμα μια φορά μας εξηγούν ότι τελικά η κλωνοποίηση δεν ε, περιλαμβάνει καμία θετική πτυχή, τουλάχιστον όχι για την ευημερία των ζώων, αλλά ούτε και για την γεωργία εν γέννη. Σίγουρα για την εκτινοτροφία την ευρωπαϊκή έτσι όπως τη γνωρίζουμε και θέλουμε να τη στηρίξουμε. Ε, έχει ήδη γίνει συζήτηση για την κλωνοποίηση εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμένα με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα το ότι συστηματικά επαναρχόμαστε ε, και κάθε φορά λέμε ότι και η κοινή γνώμη δεν είναι υπέρα όπως για τους γενετικά τροπομένους οργανισμούς. Εγώ πιστεύω πως είναι χειρότερο. Αλλά θα το μάθουμε σε λίγο γιατί θα ακούσουμε ε, τους εκπροσώπους, κάποιους εκπροσώπους ε, της κοινή γνώμη. Πάντως η κοινή γνώμη κατά με είναι πολύ λιγότερο έτοιμη να δεχτεί την κλωνοποίηση και θα έχει μια τόσο σκληρή θέση όσο αυτή που έχει και για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Γιατί επανερχόμαστε λοιπόν, ε, μάλλον επειδή υπάρχουν κάποιοι βάσιμοι λόγοι και λόγοι που δεν τους ομολογούμε πάντα. Ορισμένοι συνάδελφοι τους έχουν ήδη αναφέρει και εγώ ε, συμφωνώ με τις ανησυχίες τους. Ε, το σπέρμα το οποίο εξάγεται και οι απόγονοι που υπάρχουν σε χώρες όπως ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Αργεντινή, η και η Βραζιλία παράγουν 500.000 ε, ε, ε, τόνους κρέατος που μας έρχεται από εκεί. Εκείνες οι χώρες έχουν επιτρέψει την κλωνοποίηση. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα ανιχνευσιμότητας. Υπάρχει λοιπόν εξαπάτηση του καταναλωτή. Διερωτώ με πραγματικά γιατί <coughs> να δεχτούμε τις πρακτικές των άλλων που εφόσον δεν αντιστοιχούν στη δική μας κουλτούρα. Σας ευχαριστώ. Ο κόσμος ολόκληρος ασχολείται με το θέμα αυτό, μην το ξεχνάτε. Και μια και ο κόσμος όλος ασχολείται με αυτό το θέμα, πρέπει και εμείς να το παρακολουθήσαμε. Η κυρία Μαγκίνες. Έχετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόλις ήρθα συνάδελφοι και ζητώ συγγνώμη να σας πω τι έγινε πρόσφατα στην Ιρλανδία όπου ένα πάρα πολύ διάσημο άλογο πριν πεθάνει το 2007 ε, κλωνοποιήθηκε ε, πρόκειται για πάρα πολύ γνωστό άλογο υποδρομιών Και όταν έγινε γνωστό το γεγονός, ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί και δεν ανησυχούσε γιατί πραγματικά γνώριζαν αυτό το λόγο, το, το άλογο με συγχωρείτε, και το τι είχε επιτύχει σε διάφορες επικές επιδείξεις παγκοσμίως Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πώς έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, αν το ζώο δεν υποφέρει, όπως σε αυτή την περίπτωση που του κάναν βιοψίες, πήραν το DNA και το ζώο πέθανε. Ε, βλέπουμε πως το κοινό αντέδρασε πάρα πολύ θετικά σε αυτή την περίπτωση, καθόλου αρνητικά και ε, από την άλλη βεβαίως όταν μιλάμε για παραγωγή τροφίμων η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Θα ήθελα να ακούσω τους ειδικούς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες για, τις, ε, ε, για τα επιχειρήματά τους, αλλά ε, το επιχείρημα ότι δεν περιέχεται εδώ ο τροφικός κίνδυνος δεν ισχύει όταν βλέπουμε ότι τα ζώα αυτά πάσουν από διάφορες δυσμορφίες, παραμορφώνονται και είδαμε και έκθεση της ΕΦΣΑ για το πισμενόλ α. υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν έλεγχοι και έρευνες για την ποιότητα του κρεατός τους, σίγουρα η αντιστοιχεία στις ουσίες δεν μας επιτρέπει από μόνη της να δώσουμε θετική γνώμη. Ευχαριστώ. Δεν ζήτησε άλλος κανείς το λόγο από τους παρόντες, οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στους ομιλητές μας. Στους καλεσμένους μας. Το πολύ πέντε λεπτά στον καθένα θα ήθελα να δώσω, όχι παραπάνω και μετά στην εισηγητριά μας την κυρία Μόη. Με την ίδια σειρά που μιλήσατε και προηγουμένως. Παρακαλώ για πέντε λεπτά ο καθένας, το λόγο έχουν οι εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω το εξής. Πολλοί ευρωβουλευτές είπαν ότι οι, απόψει απόψεις δίστανται αλλά αυτό για ίσονο σημασία ζητήματα, για δευτερεύοντα. Γενικώ και εγώ και οι συνάδελφοι της Κόπα Κοζέκα έχουμε την ίδια γνώμη. Για τις επιμέρους ερωτήσεις. Ίσως εκεί που φαίνεται να διαφέρουμε είναι ως προς τα πλεονεκτήματα που ε, επιφέρει η κλωνοποίηση στην κτηνοτροφία φαίνεται ότι δεν έχει για την κτηνοτροφία ε, ωφέλη η κλωνοποίηση. Και δαπανηρή είναι και δεν είναι ούτε επωφελής βραχυπρόθεσμα. Αλλά η κλωνοποίηση γίνεται στο, προς το ανώτερο τμήμα της ε, πυραμίδας εκτροφής και αν είναι επιτυχημένη έχει απόσβεση. Βέβαια, Έχουμε πολλές δυσκολίες, λίγα πλονεκτήματα, υπάρχουν και ε, ανησυχίες για τη δημόσια υγεία. Εμείς δεν συνηγορούμε υπέρ της εισαγωγής του, της κλωνοποίησης, αλλά ε, ας μην είμαστε αφελείς και ανόητοι. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παρά τη δαπάνη, κλωνοποιούν ζώα και ίσως ε, καρπώνονται και μεγάλα ωφέλη από την κλωνοποίηση. Θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη λοιπόν. Επίσης, ε, εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μερικοί ρώτησαν αν είναι εύκολο να ανοιχνεύσουμε προϊόντα ή τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα, ώστε να μην εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτήστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ερωτήστε το Συμβούλιο. Κατά τη γνώμη μου πάντως είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε τέτοια προϊόντα. Προς το παρόν είναι μικρός ο αριθμός των κλώνων στη ΣΥΠΑ. Χρησιμοποιούνται μόνο στην κορυφή της πυραμίδας εκτροφής. Αν όμως ε, πάμε ένα βήμα παραπέρα και θέλουμε να περιορίσουμε και τους απογόνους, ε, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να απαγορεύσουμε εισαγωγές τροφίμων που θα γίνονται από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων. Και κατά τη γνώμη μου θα είναι αδύνατο να εντοπίσουμε τέτοια προϊόντα. Σκεφτείτε, έχουμε ένα τάβρο. Τον βγάζουμε από την αλυσίδα ε, διατροφής. Αν όμως έχει απογόνους, έχει γονιμοποιήσει πολλές αγελάδες και αυτό μπορεί να το κάνει ένας και μόνο τότε δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτό το κρέας πώς θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα λύσετε τέτοια προβλήματα εντοπισμού, ηχνηλασιμότητας και θεσίας Η ηχνηλασιμότητα ε, τροφίμων κλώνων μπορεί να είναι εύκολη. Αλλά η προϊόντων απογόνων κλώνων αυτή είναι σχεδόν αδύνατη. Και αυτό θα είναι το μέτρο με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Μάλλον θα διαβάσετε τα έγγραφα που κυκλοφορούν από την αντίστοιχη υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν ξέρω αν θέλουν να συνεργαστούν ή να καταλήξουν συμφωνία με τους Ευρωπαίους. Πάντως ε, για το θέμα αυτό μάλλον θα ήταν διστακτική και απρόθυμη. Ρωτήσατε γιατί συνεχίζουμε την έρευνα. Γενικώ. Και αν όλο ο κόσμο δεν ε, ασχολούνται με, με την κλωνοποίηση, ούτε και εμεί θα θέλαμε να κλωνοποιήσουμε. Αλλά ζούμε στο σύγχρονο κόσμο και θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε μια κτηνοτροφία που δεν περιορίζεται μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, αλλά είναι γενική. Και πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και απέναντι στον Καναδά και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και η ποσότητα σπέρματος που εξάγουν οι χώρες αυτές είναι δεκαπλάσια από αυτή που εξάγουμε εμείς. Οπότε είναι πολύ δύσκολος, σκληρός ο ανταγωνισμός με τον Καναδά και τη ΣΥΠΑ. Και αν έχουν τύχει να εκθρέψουμε, ε, αν εκθρέψουν ε, κλωνοποιημένο τάβρο πολύ καλύτερο από ό,τι εμείς, τότε εμείς έχουμε χάσει τον ανταγωνισμό. Και τώρα, σε ό,τι είπε ο Δόκτωρ Μπρούμ. Εμείς ε, δεν εκτρέφουμε για γαλακτοπαραγωγή. Μέχρι το 2000 το κάναμε θέλαμε περισσότερο γάλα, περισσότερο λίπος, περισσότερη πρωτεΐνη. Αλλά από το 2000 και μετά έχουμε αλλάξει την κατεύθυνση. Μας ενδιαφέρει η μακροζωία, η υγεία και αναπαράγουμε ή εκτρέφουμε γελάδες που θέλουμε να παραμείνουν στη φάρμα για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Γιατί αλλάζουν οι συνθήκες συνεχώς. Έχουμε τις κλιματικές αλλαγές για παράδειγμα και εμείς προσαρμοζόμαστε και αλλάζουμε τις συνήθειες και τους τρόπους εκτροφής και ίσως από αυτήν την άποψη κλωνοποίηση θα μπορούσε να βοηθήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ε, εμπειρογνώμονος, ο κύριος Νταβίτ. Παρακαλώ, πέντε λεπτά το πολύ. Εγώ θα μιλήσω αγγλικά και να με συγχωρείτε κύριε Φεράν γιατί εκπροσωπώ την Κόπα Κοσέκα μια ευρωπαϊκή οργάνωση και παρά το ότι βεβαίω είμαι μεγάλος και περήφανος γι' αυτό ε, εργαζόμαστε στα αγγλικά και εγώ θεωρώ πως η Ευρώπη είναι η καλύτερη ευκαιρία της γαλλικής γλώσσας. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε παρακάτω. Τώρα, κυρία Αγγιλέρα, θα ήθελα να επανέλθω στην παρατήρησή σας Ε, θα προτιμούσαμε λοιπόν εμείς ε, έναν κανονισμό παρά μια οδηγία για να είμαστε σίγουροι ότι θα εφαρμοστούν τα ίδια πράγματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα θα σας δώσω το παράδειγμα της πρότασης που συζητιέται αυτή τη στιγμή στην Κομισιόν για έναν κανονισμό με στόχο να αντικαταστήσει μια, πρώην, μια παλιά οδηγία που είχε εφαρμοστεί με τελείως διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα. Γι' αυτό αν είναι να ε, νομοθετήσετε καλό θα είναι να είναι κανονισμός ε, για να μην έχουμε πρόβλημα ε, με τη διαφορετική εφαρμογή ειδικά για την ιχνηλασιμότητα. Κατόπιν για το σχόλιο του κυρίου Μποβέ συμφωνώ μαζί του πλήρως. Δεν χρειάζεται ε, κλωνοποίηση για να έχουμε ε, βιώσιμη κτηνοτροφία. Η Ευρώπη έχει την δυνατότητα ε, να έχει μια, ένα αναλλακτικό μοντέλο σε σχέση με τη ΣΥΠΑ και την Κίνα. Ε, οι ΙΠΑ προτείνουν δύο προτεραιότητες ράτσα, Χολστάιν για γαλακτοκομικά και Άγκους για κρέας. Στην Ευρώπη για γάλα έχουμε και Μομπελιάρα και τις σκανδιναβικές κόκκινες ράτσες, Νορμάν και άλλες. Για κρέας, πέρα από την Άγκους που είναι μία ράτσα, έχουμε και άλλες ράτσες ε, και από τη Γαλλία, την Ιταλία και Ανατολική Ευρώπη κτλ. Οπότε ναι, η γενετική ε, ποικιλία είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ε, κτηνοτροφίας και εντός της κάθε ράτσας και όσον αφορά τη, τις πολλές ράτσες. Και συμφωνώ λοιπόν μαζί σας πλήρως και θεωρώ πως ε, είναι ε, μαζί σας εδώ πέρα ο κλάδος και αυτό θα ωφελήσει την ποικιλία τη γενετική. Κάτι άλλο. Εντάξει, ναι, υπάρχει Ευρώπη, υπάρχει απέτηση της κοινωνίας, δεν χρειάζεται να... Ε, δεν, ε, αποδέχεται ο κόσμος την εμπορία ε, τροφίμων από κλόνους, όλοι συμφωνούν με αυτό, αλλά είμαστε σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο με εισαγωγές όχι μόνο σπέρματος και εμβρίων αλλά και τροφίμων. Και πρέπει να γνωρίζουμε πώς. Χωρίς ίχνη λασιμότητα στα σύνορα ή διαφάνεια από τους εισαγωγείς και όχι μόνο για την καταγωγή αλλά και στο τι γίνεται με κάθε ε, ζώο που εισάγεται για αναπαραγωγή, ε, δεν θα φτάσουμε πουθενά. Γιατί με το DNA δεν βρίσκουμε άκρη. Το DNA κλόνου και μη είναι το ίδιο. Θα πρέπει στην καταγωγή ε, να λένε πως πρόκειται για κλόνο του ζώου αυτού. Αυτά είναι τα τρία μου σχόλια για τις ε, ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που κάνατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο καθηγητής ο κύριος Μπρούμ για πέντε λεπτά. Thank you. Uh, firstly, there was, uh, there were questions... Ευχαριστώ. Υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις ε, που έλεγαν γιατί χρειαζόμαστε την κλωνοποίηση. Νομίζω απαντήθηκε από τον κύριο Φένεμαν. Επίσης να πούμε πως ένας από τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε την κλωνοποίηση είναι να διονύσουμε γενετικά τροποιημένες γραμμές σε άλλα μέρη του κόσμου. Ε, γίνεται αυτό και ε, για την έρευνα στην Ευρώπη όταν έχουμε ένα γενετικά τροποποιημένο ζώο, χρησιμοποιούμε ε, κλωνοποίηση και νομίζω θα διαδοθεί αυτό στο μέλλον. Κάτι άλλο. Μου απευθύνθηκε μια ερώτηση από την κυρία Χάνσεκαμπ για το αν είχαμε βελτιώσει στην τεχνική όσον αφορά τις ε, δυσκολίες ε, στο να γεννήσουν οι μητέρες και όσον αφορά τις δυσμορφίες ε, στα ζώα. Η απάντηση είναι πως ε, υπάρχει κλωνοποίηση εδώ και πολύ καιρό, αλλά στα θηλαστικά οι μέθοδοι πλέον αυτές ε, χρησιμοποιούνται εδώ και 16 χρόνια και έχουμε λίγο πολύ τα ίδια προβλήματα. Οπότε δεν έχει υπάρξει σοβαρή βελτίωση και δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα βραχυπρόθεσμα. Τώρα, μιλώντας για διαφορετικά είδη, σας έδωσα κάποιες απαντήσεις. Ε, υπάρχουν προβλήματα πράγματι για τις μητέρες, τα θηλαστικά και για τους απογόνους ε, σε, σε θηλαστικά πτηνά και ψάρια, σε όλα τα ζώα δηλαδή. Και στα άλογα, επειδή αναφέρθηκε μια Ιρλανδή βουλευτής σε ένα άλογο. Αν κλωνοποιήσετε άλογο και αυτό πρόβλημα θα έχει δεν έχει γίνει ε, σοβαρή έρευνα, αλλά δεν βλέπω λόγο γιατί να μην αντιμετωπίζει και το άλογο το ίδιο πρόβλημα. για το τι γίνεται σε άλλες ε, χώρες. Ε, γεγονός είναι πως σε άλλες χώρες ο κόσμος δεν ανησυχεί τόσο το κοινό για τα ζητήματα αυτά της ευζοίας των ζώων και επιτρέπεται σε ιπα Αργεντινή και κάνα δύο χώρες ακόμα γιατί αγνοούν αυτή την πτυχή ε, κάτι το οποίο το ευρωπαϊκό κοινό δεν ανέχεται να ταλαιπωρούνται δηλαδή έτσι τα ζώα. Ε, οι άλλες χώρες δεν το βλέπουν έτσι, αν και υπάρχουν κάποια σημάδια ότι κινούνται προς τα εκεί. Μετά, το ζήτημα είναι αν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τα ζώα, πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε διαβατήρια για τα βοηδή, ε, υπάρχει η χνηλασιμότητα. Έχουμε τσιπάκια στα ζώα, τα ταυτοποιούμε με το DNA τους και στο προσεχές μέλλον θα μπορούμε να ταυτοποιούμε τα ζώα με τρόπο πολύ φτηνότερο μέσω του DNA, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ε, αρκετά ακριβό. Αλλά σε λίγα χρόνια θα αλλάξει. Αν μπορούμε λοιπόν να ταυτοποιήσουμε ζώα που είναι απόγονοι ε, κλωνοποιημένων ζώων ή από εισαγόμενο σπέρμα και εισαγόμενα οάρια. Η απάντηση είναι ότι πρέπει να μας δώσει τα αρχεία ο προμηθευτής. Ε, εάν είναι λοιπόν ειλικρινείς οι προμηθευτές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αρχεία όπως τα χρησιμοποιούμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την σήμανση των ζώων. Αλλά όπως είπε ο κύριος Νταβίδ δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε απολύτως ένα ζώο ως κλόνο ή απόγονο κλόνο, δεύτερη ή τρίτη γενιά, ε, από το DNA. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο αρχείο και μετά να το συσχετίσουμε με κάποιες πληροφορίες που έχουμε για το DNA των ε, γονέων. Υπάρχουν δυνατότητες αλλά θα κοστίζει. Ε, μιλάμε για πάρα πολύ μικρό αριθμό ζώων ε, που εισάγονται. Πόσα δείγματα σπέρματος, πόσα οάρια εισάγονται. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Όλα αυτά λοιπόν, το κάθε ένα θα πρέπει να έχει ένα πλήρες αρχείο του από πού προήλθε το σπέρμα. Ε, κάτι το οποίο ήδη απαιτείται, οπότε δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι εφόσον τηρείται αρχείο, αν είναι εκλονοποιημένο δεν θα το φέρετε. Αλλιώς το κοινό θα, θα αρνηθεί. Δεν είναι δυνατόν να τα απαγορεύουμε στην Ευρώπη αλλά να το επιτρέπουμε εισαγόμενο. Εάν μπορούμε λοιπόν να το ταυτοποιήσουμε, καλό θα είναι και νομίζω πως θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε με τις απαντήσεις. Ευχαριστώ θερμά τους ε, εμπειρογνώμονες και μετά την ολοκλήρωση του πρώτου πάνελ θα δώσω το λόγο στην, μας, στην εισηγητριά μας, συγγνώμη, την κυρία Μόη. Εγώ ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση στον καθηγητή Μπρούμ και ακολουθώ το πρόγραμμα όπως το έχουμε προκαθορίσει, αν θέλετε. Πολύ σύντομα έχουμε ελάχιστο χρόνο, αλλά προλαβαίνετε μια ερώτηση. Μια απλή ερώτηση θέλω να υποβάλω έπειτα τα συμπεράσματα μετά μαζί με τη συνάδελφο Ζόμερ. Ε, ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή Μπρούμ όσον αφορά την υγεία των ζώων. Είδαμε από μελέτε ότι αυτά τα ζώα τα κλωνοποιημένα και οι μητέρε επίση πρέπει να ε, να ε, καταναλώσουν μεγάλες ποσότητες ορμονών. Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι αυτές οι ορμάνες δεν θα περάσουν ε, στους πολίτες μας από τη στιγμή που καταναλώνουν το κρέας αυτών των ζώων με ορμόνες. Και αυτό η υψηλή τα υψηλά ποσοστά ορμονών δεν τροποποιούν τα κύτταρα των απογόνων και δεν οδηγούν εν πάση περιπτώσει σε αλλαγές ε, στη βιοσύνθεση ή στα κύτταρα των απογόνων που συνήθως ε, οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές. Θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν τέτοιο είδους μελέτες ε, και για τα ζώα. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, κύριε Μπρούμ, πώς θα μπορούσατε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Αναφέρθηκε από τον κύριο Μποβέ ότι η χρήση ορμονών, η ορμονοθεραπεία στη διαδικασία θα επηρεάσει τις συνθήκες διαβίωσης της μητέρας, την ευημερία της μητέρας. Όντως, εκεί βλέπουμε αρνητικά αποτελέσματα από την ορμονοθεραπεία. Εσείς όμως μιλήσατε για τις επόμενες γενιές. Αν χρησιμοποιεί κανείς ορμόνες για την αναπαραγωγή των μητέρων που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή κλώνων, δεν βλέπω γιατί να επηρεάζονται οι απόγονοι, οι επόμενες γενιές. Οι ορμόνες που παίρνει η μητέρα δεν θα επηρεάσουν τις επόμενες γενιές. Θα επηρεάσουν μόνο την μητέρα. Ίσως και την ευημερία του νεογνού. Αλλά εκεί σταματά η αρνητική συνέπεια στην ευημερία. Όχι, δεν επεκτείνεται στις ε, επόμενες γενιές. Ε, δεν κατάλαβα αν μπορούμε να ελέγξουμε το επίπεδο της, της ε, υγειονομικής ε, επιθεώρησης. η Κομισιόν. Ε, κάποιες ερωτήσει απευθύνθηκαν προς την Κομισιόν και εν μέρει απάντησαν οι πυρογνώμονες, αλλά και εγώ αισθάνομαι υποχρέωση να απαντήσω. Καταρχήν, είπατε πως πιέζει η Κομισιόν ξανά και ξανά για την κλωνοποίηση. Πιστεύω πως δεν είναι σωστή αυτή η αντίληψη. Το θέμα είναι πως υπήρξε μεγάλη ζήτηση, πολύ έντονο το αίτημα από το Κοινοβούλιο να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Και αυτό που έχετε επιτάπητος είναι η ανταπόκρισή μας σε αυτό το αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη την θέση και του ευρωπαϊκού κοινού που θέλει το ζήτημα, ζήτημα αυτό να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να θυμίσω ότι αυτό που προτείνουμε είναι απαγόρευση των κλώνων και των τροφίμων από, που προέρχονται από κλόνους. Εγώ αυτό που άκουσα ως συζήτηση σήμερα αφορά τους απογόνους, γιατί κατά τα λοιπά συμφωνούμε. Ε, η πρόταση αντιποκατοπτρίζει τα όσα υπόθηκαν εδώ στην αίθουσα από, σχεδόν, από πολλούς ε, το θέμα είναι λοιπόν τι κάνουμε με τους απογόνους, με τις επόμενες γενναίες. Και εδώ να θυμίσω ότι καταρχήν η μελέτη γίνεται, αλλά, οι μελέτες μάλλον συνεχίζονται, αλλά πραγματικά δεν έχουμε καμία επιστημονική μέθοδο για να διακρίνουμε τα τρόφιμα γάλα, προϊόντα γάλακτος ή κρέατα από τους κλόνους, που προέρχονται από κλόνους, από τα υπόλοιπα δεν υπάρχει κανένα απολύτω εργαλείο. Όπως είπαν οι εμπειρογνώμονε, ο μόνος τρόπος είναι διοικητικό. Δηλαδή να υπάρχει μια γνηλασιμότητα ε, γραπτή που θα πηγαίνει πίσω δεν ξέρω πόσες γενιές. Επίσης θα έπρεπε να σκεφτούμε και άλλο ένα στοιχείο. Υπάρχουν κάποιες, αλλά υπάρχουν εισαγωγέ. Ε, ε, σπέρματος ή οαρίων από τις χώρες όπου επιτρέπεται η κλωνοποίηση και θέλω να ρωτήσω τους Ευρωπαίους κτηνοτρόφους και γεωργούς αγρότες γιατί θέλουν να εισάγουν αυτό το είδος το ε, σπέρμα. Συνήθως πρόκειται για υψηλή ποιότητας ζώα που αντιπροσωπεύονται από αυτό το γενικό, γενετικό υλικό. Αν πρέπει όμως να διακρίνουμε ανάμεσα στους κλώνους και τους μη κλόνους και ε, ε, απαγορεύουμε όλες τις εισαγωγές συμπεριλαμβανομένου και του πολυαποδοτικού σπέρματος που μπορεί να χρειάζεται στην κτηνοτροφία στην Ευρώπη. Συμφωνώ ότι στο κλωνοποιημένο οάριο ή σπέρμα ίσως να είναι ευκολότερο να βρεθεί η λύση με την, με την ακόμα και αν είναι διοικητικού τύπου ε, ε, ε, για τους απογόνους όπου υπάρχει πρόβλημα και μεγάλος αντίκτυπος, όπου πιστεύω μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε επίσης προβεί στην αξιολόγησή μας. Ωραία, ολοκληρώνουμε το πρώτο πάνελ και σας ευχαριστώ θερμά. Έχουμε ολιγόλεπτη καθυστέρηση και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό από τον συμπρόεδρο Λαβία, στον οποίο δίνω και τη σκητάλη για την Προεδρία του επόμενου πάνελ. Ευχαριστώ κύριε Σεκέρσκι. Περνάμε στο δεύτερο πάνελ της Δημόσιας Ακρόασης. Θα πραγματευτούμε θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δηλαδή κυρίως ε, τα επιστημονικά και διδεολογικά ε, θέματα, τις πτυχές αυτές, ε, καθώς και την προοπτική των καταναλωτών. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια της Επιτροπής ΕΜΒΗ, την κυρία Σόμερ, για να μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή και μετά θα ακούσουμε τους τρεις καλεσμένους μας. Κυρία Σόμερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με ενδιαφέρον ε, τους ομιλητές από το πρώτο πάνελ. Ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπαν και περνάμε τώρα στο δεύτερο πάνελ το κομμάτι δηλαδή της Επιτροπής Περιβάλλοντος, τις επιστημονικές και δεοντολογικές πτυχές ε, της κοπιά των καταναλωτών. Χαίρομαι που έχουμε ομιλητές υψηλού επίπεδου, κάποιον από την ΕΦΣΑ, μάλιστα από το τμήμα επιστημονικής στρατηγικής τον κύριο Ρόμπινσον μετά κάποιον από την Ευρωπαϊκή Ομάδα για την Δεοντολογία της Επιστήμης που παίζει βεβαίω σημαντικό ρόλο και τέλος μια εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών για να συζητήσουμε ακριβώς ε, το θέμα αυτό και την σκοπιά ε, των ε, καταναλωτών. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για... αναμένομη αγωνία δε το δεύτερο μέρος συζήτησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο έχει ο κύριος Τόμπιν Ρόμπινσον προϊστάμενο του τμήματο επιστημονική στρατηγική και συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων για μια παρουσίαση 10 λεπτών. Κατόπιν ετήματο τη ε, Κομισιόν η ΕΦΣΑ υιοθέτησε μια γνωμοδότηση τον Ιούλιο του 2008 για το θέμα και έγιναν περαιτέρω δηλώσεις το 2009 και 2010 το τμήμα του κυρίου Ρόμπινσον είναι υπεύθυνο για το θέμα αυτό, είπαμε, της επιστημονικής στρατηγικής και συντονισμού, αλλά και για τους νέους κινδύνους στην ε, διατροφική αλυσίδα. Κύριε Ρόμπινσον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να συνεψίσω την δουλειά που κάνουμε στην ΕΦΣΑ για το θέμα αυτό. Θα ξεκινήσω υπενθυμίζοντάς σας τον ρόλο της υπηρεσίας μας. Είναι, θα έλεγα, θεμέλιος λήθος της αξιολόγησης κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ασφάλεια των τροφίμων. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και σε ανοιχτή διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους και βεβαίω υπάρχουμε για να δίνουμε σε εσά ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές ε, και σαφή, σαφείς ε, οδηγίες για τον κίνδυνο που υπάρχει και πιθανούς μελλοντικού κινδύνους. Ε, δρούμε ανεξάρτητα από την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη και χρηματοδοτούμαστε βεβαίως από τον Ευρωπαϊκό Προεπλογισμό. Στο συγκεκριμένο θέμα μας έχουμε λάβει αρκετές ερωτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ζητούν μια επιστημονική γνωμοδότηση για, ζήτημα, για το ζήτημα της ασφάλειας τροφίμων, της υγείας των ζώων και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δώσαμε επιστημονική γνωμοδότηση τέσσερις φορές το 2008, 2009, 2010 και 2012 και Πρόκειται για επιστημονική γνωμοδότηση για να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή η οποία διαχειρίζεται το πέρα κίνδυνο. Η επιστημονική γνωμοδότηση του 2008, όπως είπαμε, ήταν κατόπιν ετήματος της Επιτροπής Υπήρξε μια δημόσια διαβούλευση, όλοι είχαν την ευκαιρία να συνεισφέρουν. Ε, λάβαμε συνεισφορές από 68 διαφορετικούς φορείς. Ε, τα συμπεράσματα ήταν πώς. Στον τομέα της κλωνοποίησης το 2008 είχαμε επαρκή δεδομένα, περιορισμένα μόνο, για χείρους και βοηδοί. Ξέραμε τα προβλήματα στα ανήλικα άτομα και δεν υπήρχαν ε, ανησυχίες ασφάλειας τροφίμων για το κρέας και το γάλα από τα ζώα αυτά. Το 2009 και πάλι η Κομισιόν ζήτησε μια επικαιροποίηση της γνωμοδότησης αυτής με ειδικό βάρος στην υγεία των ζώων αυτών και επίσης με ένα συγκεκριμένο ερώτημα εάν είναι δυνατόν να ε, προχωρήσουμε και στην αξιολόγηση για τα εγωπρόβατα και τα πουλερικά. Και επαναβεβαιώσαμε τα συμπεράσματα του 2008 και είπαμε πως δεν ήταν δυνατόν να γίνει επέκταση για άλλα είδη με τα τότε υπάρχοντα δεδομένα. 2012 και πάλι μας ζητήθηκε μια επικαιροποίηση με ακριβώ τα ίδια ερωτήματα Συγκεκριμένα το 10 και 12 αναθεωρήσαμε πλήρως την βιβλιογραφία και είχαμε πάλι μια ανοιχτή πρόσκληση για δεδομένα σε οποιονδήποτε ήθελε να συνεισφέρει στις ε, συζητήσεις ε, που έκαναν οι ειδικοί μας και πάλι το 10 και 12 επαναβεβαιώσαμε τα συμπεράσματα των ε, προηγούμενων δηλώσεων. Ποια ήταν λοιπόν αυτά τα συμπεράσματα στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων από τις μελέτες που είχαμε. Δεν είδαμε διαφορές ε, όσον αφορά την σύσταση των ε, τροφίμων, κρέατος και γάλακτος ε, από υγιή συμβατικά ζώα. Μιλάμε για αμπινοξέα, βιταμίνες, ασβέστιο, περιεχόμενο σε περιεκτικότητα σε νερό ήταν ταυτόσιμα με μη κλωνοποιημένα ζώα. Το ίδιο όσον ε, αφορά και άλλους ε, παράγοντες, όμως πρέπει να σημειώσουμε πως δεν υπάρχουν μακροχρόνιες μελένες ε, τοξικότητας, μάλλον γιατί δεν υπάρχει και το ανάλογο κίνητρο. στον τομέα της υγείας και της ευζοίας των ζώων. Τα ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές. Έχουμε πρώτα απ' όλα αυξημένο αριθμό θανάτων σε όλες τις φάσεις από το έμβριο μέχρι τα ανήλικα άτομα. Και βεβαίως είχαμε και ανώμαλη τοποθέτηση του πλακούντα που οδηγούσε συχνά σε θανάτους εμβρίων. Και, υπήρχε βέβαιος, και υπήρχαν και επιγενετικές δυσλειτουργίες και οι ανησυχίες αυτές βεβαίω δεν επηρεάζουν ε, τους απογόνους των κλώνων ε, που αναπαράγονται με τρόπο συμβατικό. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της κλωνοποίησης, το είπαν και άλλοι ομιλητές, υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις ε, στην έρευνα, αλλά είναι μικρές. Δεν υπάρχει ουσιαστική βελτίωση της ε, αποτελεσματικότητας ε, της κλωνοποίησης. Για γελάδες ε, το ποστό επιτυχίας κλωνοποίησης είναι μεταξύ 6 και 15% ε, ενώ η τεχνητή κονομοποίηση μη κλωνοποιημένων ζώων ε, είναι 45 με 60% για τα κουρούνια, δε το ποστό επιτυχίας κλωνοποίησης κυμαίνεται γύρω στο 6%. Τέλος, το τελευταίο ερώτημα αφορούσε τους ε, κινδύνους για το περιβάλλον και, και στις τέσσερις αξιολογήσεις ε, δεν είδαμε κινδύνους για την γενετική ποικιλία ή την βιοποικιλότητα του περιβάλλοντος. Με τα δεδομένα λοιπόν που υπάρχουν δεν φαίνονται κάποιοι δείκτες οι οποίοι δείχνουν πως προκύπτουν νέοι επιπρόσθετοι κίνδυνοι από τα κλωνοποιημένα ζώα σε σύγκριση με τα συμβατικά. Καμία πληροφορία που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν ε, μας λέει πως μπορούμε να φοβόμαστε, πως υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Και εδώ πέρα τελειώνω και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στον επόμενο μας ε, καλεσμένο εμπειρογνώμονα, τον κύριο Πέρε Πουγκντομενέκ Ρόσελ, από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Δεοντολογίας στην Επιστήμη και τις Νέες Τεχνολογίες. Θα μας κάνει μια δεκάλεπτη παρουσίαση σε σχέση με την γνωμοδότηση της ε, Ευρωπαϊκής Ομάδας Δεοντολογίας στην Επιστήμη και τις Νέες Τεχνολογίες. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ομάδα Δεοντολογίας στην Επιστήμη και τις Νέες Τεχνολογίες έλαβε στα τέλη του 2007 έτοιμα από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια γνωμοδότηση των δεοντολογικών πτυχών της κλωνοποίησης των ζώων που σχετίζονται με την παραγωγή τροφίμων. Η γνωμοδότηση δημοσιεύθηκε και μπορείτε να τη βρείτε Οπότε σας παραπέμπω και για τις λεπτομέρειες. Αυτό που είπε η ομάδα μετά τη λήψη του αιτήματο από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να οργανώσει μία δημόσια κρόση με εμπειρογνώμονες. Δηλαδή εμπειρογνώμονες, επιστήμονες αλλά και εκπροσώπους των κτηνοτρόφων ε, για να συλλέξουμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Επίσης, ε, οργανώσαμε και δημόσιες διαβουλεύσεις για το θέμα αυτό, από τις πρώτες και όλα. Λάβαμε πάνω από 300 ε, απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που στείλαμε για τις διαβουλεύσεις. Οργανώσαμε και ένα στρογγυλό τραπέζι στις Βρυξέλλες με διαφερόμενους από πολλές πλευρές που μας παρουσίασαν, ένα ευρύ φάσμα απόψεων και με όλα αυτά τα στοιχεία εκπονήσαμε μια γνωμοδότηση που στην ουσία συνοψίζει όλες αυτές τις ε, θέσεις, ε, κάνει μια συμπίλησή τους και προβαίνει σε κάποιες συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα βασικά δεντολογικά προβλήματα που εγείρει το θέμα της κλωνοποίησης. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε καταρχήν τις ε, δεοντολογικές ανησυχίες και προβληματισμούς για το θέμα αυτό και διαιρέσαμε τη γνωμοδότησή μας σε τέσσερα κεφάλαια. Το ε, πρώτο αφορά τα ίδια τα κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους. Από εκεί και πέρα ε, διαπιστώσαμε ότι πολλοί, όπως είπατε και εσείς, ε, ανησυχούν με την αυξανόμενη χρήση ε, των ζώων για τέτοιους σκοπούς. Ε, προβληματίζονται με τη, για την ακεραιότητα των ζώων, τα δικαιώματά τους, την υγεία των ζώων, αλλά και την ευημερία των ζώων, τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν ανησυχίες και για την ανθρώπινη υγεία. την ανθρώπινη υγεία και την ε, ανθρώπινη ευεξία, την ασφάλεια αλλά και την προστασία των ανθρώπων. σε σχέση με τα επιχειρήματα της τεχνολογίας ε, σε περίπτωση που αφορά παράγωγη τροφίμων. Οπότε ο προβληματισμός για την ε, επιστηστική ασφάλεια είναι σημαντικός. Επίσης μας απασχόλησε το θέμα μήπως γίνει κατάχρηση βάρος των ανθρώπων αν δεχτούμε την κλωνοποίηση των ζώων, θα μπορούσαμε να ολιστήσουμε και προς την αποδοχή της ίδιας τεχνολογίας για κλωνοποίηση των ανθρώπων. Κάτι που απογοητεύεται, απογορεύεται συγγνώμη, πλήρως σε όλες τις χώρες η κλωνοποίηση των ανθρώπων. Άλλος προβληματισμός αφορούσε το περιβάλλον. Το θέμα της γενετικής πολυμορφίας που θέλουμε να διαφυλαχθεί, της γενετικής πολυμορφίας των ειδών. Επίσης το θέμα της βιοασφάλειας και της ε, περιβαλλοντικής αηφορίας, ε, της ρήπανσης ε, ή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η αυξανόμενη χρήση κάποιων ειδών για την κρεατοπαραγωγή ίσως δημιουργήσει προβλήματα σε όλους τους παραπάνω πλάτους. Και κάποιος προβληματισμός και ανησυχίες για την ίδια την κοινωνία πώς το κοινό αντιλαμβάνεται αυτά τα θέματα, πώς, αν υπάρχει αποδοχή της κλωνοποίησης ε, ή τι γίνεται με τους καταναλωτές, ποια είναι η θέση των καταναλωτών. Οπότε αναλύσαμε όλα αυτά τα θέματα και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν διαφορές, διαστάσεις απόψεων. Και υπάρχουν και κάποια προβλήματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα και την βιομηχανοποίηση, την αηφορία της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Όλα αυτά τα θέματα βέβαια δεν είναι ειδικά θέματα της κλωνοποίησης. Είναι γενικότερα θέματα που προβληματίζουν τους χρήστες, τους καταναλωτές των γεωργικών προϊόντων και των κτηνοτροφικών προϊόντων. Τα οι βασικοί προβληματισμοί, οι βασικές αφορούσαν την ευημερία των ζώων, την επιστημιστική ασφάλεια, την ασφάλεια των τροφίμων, την πολυμορφία και την αντίληψη που έχει το κοινό για τα θέματα αυτά. Τώρα, γιατί χρησιμοποιούνται αυτές οι τεχνολογίες και εγείρουν προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δικαιώματα στις τεχνολογίες αυτές, οπότε μπορούν να απαιτήσουν διπλώματα τεχνίας, γιατί μπορεί να έχουν περιορισμένη επιτυχία αυτές οι τεχνικές, αλλά έχουν κάποια επιτυχία, οπότε δημιουργούν και πνευματικά δικαιώματα. Μπορεί αυτό το ζήτημα προς το παρόν είναι περιθωριακό, αλλά υπάρχει. Το μείζον ζήτημα αφορά την ασφάλεια των τροφίμων φυσικά. την εποχή που ετοιμάζαμε τη γνωμοδότηση, λάβαμε την πολύ διεξοδική γνωμοδότηση της Αμερικανικής Φαρμάκων και Τροφίμων. Πολύ εμπεριστατωμένη έκθεση, πληρέστατη και μεστή. Επίσης ε, είχαμε και τις ε, γνωμοδοτήσεις τη ΕΦΣΑ που σε μεγάλο βαθμό συμπίπτουν με, τις, με τη γνωμοδότηση της Αμερικανικής Υπηρεσίας ε, Τροφίμων και Φαρμάκων. Γιατί τα ίδια τα κλωνοποιημένα ζώα δεν θα εισέλθουν στην ε, αγορά τροφίμων. Πρόκειται για πολύ ακριβά τα πανηρά ζώα. Αυτά που θα εισέλθουν στην αγορά είναι οι απόγονοι αυτών των κλωνοποιημένων ζώων. Και όλες οι εκθέσεις που εξετάσαμε καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν δημιουργούν οι απόγονοι κλωνοποιημένων ζώων ε, ανησυχίες ε, για τη δημόσια υγεία. Αν υπήρχαν τέτοιες ανησυχίες δεν θα χρησιμοποιούνταν τέτοια ζώα. Αυτό το, το επιχείρημα γίνεται αποδεκτό. Αλλά υπάρχει πρόβλημα με την ευημερία των ζώων. Αυτή εξακολουθεί να δημιουργεί προβληματισμό γιατί ισχύει ότι η αντίληψη που επικρατεί στην Ευρώπη για την ευημερία των ζώων είναι διαφορετική από την αντίληψη σε άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Λατινική Αμερική. Και αυτό το πρόβλημα παραμένει, η διαφορά αντίληψης. Και δεν το έχουν λύσει οι νέες τεχνολογίες. Άλλο ζήτημα προκύπτει με την πολυμορφία, τη γενετική πολυμορφία. Η κλωνοποίηση περιορίζει τη γενετική πολυμορφία των ε, ζώων εκτροφής. Αυτό ισχύει βέβαια και για τα φυτά που κλωνοποιούνται. Αλλά η κλωνοποίηση είναι μια ακραία περίπτωση περιορισμού της ε, γενετικής πολυμορφίας. Θα μπορούσατε να πείτε ότι αυτό το κάνουμε και με τις ε, συνηθισμένες πρακτικές. Πριν από ένα μήνα ένας, ε, πέθανε ένας μη κλωνοποιημένος ε, τάβρος με 500.000 απογόνους. Οπότε είναι μια τάση μείωσης της γενετικής πολυμορφίας ε, και με τις κανονικές μεθόδους, χωρίς καν κλωνοποίηση. Αλλά αυτή η μείωση της γενετικής πολυμορφίας ανησυχεί την κοινή γνώμη μπορούσε να πει κανείς ότι σε μερικέ περιπτώσεις η κλωνοποίηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να προστατευτούν ή διαφυλαχθούν είδη που βρίσκονται στο χείλος της εξαφάνισης. Και αυτό ισχύει, αλλά και αυτό είναι δευτερεύον προς το παρόν. Και τέλο, η αντίληψη του κοινού. Η αποδοχή της κλωνοποίηση ε, στην κοινή γνώμη. Αυτό το ακούσαμε και προηγουμένως. Γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να καταλήξει σε μια δημοσκόπηση μέσω του Ευρωβαρομέτρου που έγινε πολύ γρήγορα και δημοσιεύθηκε στα τέλη του 2008 και μάλιστα το Ευρωβαρόμετρο η δημοσκόπηση αυτή επιβεβαίωσε τις δικές μας ιδέες. Τώρα, εν κατακλείδη, για τα θέματα ευημερίας των ζώων, ευεξίας ή καλών συνθηκών διαβίωσης, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ε, υπάρχει θέμα αναλογικότητας εδώ, γιατί υπάρχει διαφορά με την κλωνοποίηση για παραγωγή τροφής. Είναι περιορισμένα σίγουρα τα ωφέλη σε σχέση με την ευημερία και την κοινωνική αποδοχή. Συζητήσαμε και το θέμα της ετικετοθεσίας της σήμανσης. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι τεχνικά να βάλουμε ετικέτες στα προϊόντα αυτά. Σκεφτείτε, αν έχουμε ένα λουκάνικο που έχει υπεραχθεί από κρέας πολλών και διαφορετικό ζώο, τι ετικέτα να βάλουμε ή το ίδιο ισχύει για το γάλα. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Και για το DNA, ούτε οι τεχνικές DNA θα μας βοηθήσουν να λύσουμε το πρόβλημα της ετικετοθεσίας. Εκτός αν ε, εξελιχθούν πολύ Προς το παρόν όμως δεν έχουμε τόσο προηγμένες τεχνικές DNA. Οπότε ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει όλες αυτές τις πτυχές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Καμίγε Πεγά που είναι προϊστάμενη στο ΜΠΕΟΚ που είναι Ευρωπαϊκός Οργανισμός, Οργάνωση μάλλον των Καταναλωτών και θα μας μιλήσει για την ε, γνώμη των καταναλωτών για το θέμα της κλωνοποίησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε αυτή την ακρόαση ακούσαμε ήδη διάφορες πτυχές ε, της κλωνοποίησης και αυτή τη στιγμή θα ήθελα εγώ να σας παρουσιάσω την άποψη των Ευρωπαίων καταναλωτών όσον αφορά της, ε, την κλωνοποίηση για την παραγωγή τροφίμων. Θα στραφώ άμεσα στην στάση των Ευρωπαίων προς την κλωνοποίηση των ζώων. Όπως ο προηγούμενος ομιλητής είπε, ε, έχει αυτό, ε, έχουν γίνει δύο σφυγμομετρήσεις σε δύο έρευνες του Ευρωβαρόμετρου το 2008 και το 2010 και στις δύο οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ήταν κατά ε, το της κλωνοποίησης για την ε, παραγωγή τροφίμων. Είχαν ανησυχίες ε, για τα μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλωνοποίησης στην φύση. Θεωρούν πως είναι πλήρως ε, απαράδεκτη για την ε, παραγωγή τροφίμων. Τα δύο τρίτα συμφωνούν ότι υπάρχουν ηθικοί λόγοι για την απόρριψη της κλωνοποίησης των ζώων και 83% είπαν ότι θα ήθελαν τα τρόφιμα από κλόνους ή από γόνους αυτών να, ε, είναι, να φέρουν ετικέτες εάν ε, προωθηθούν στα ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ. Οι Αμερικανοί καταναλωτές επίσης δείχνουν παρόμοιες ανησυχίες και δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι 53% των Αμερικανών δεν είναι πιθανό να αγοράσουν ε, κρέας, γάλα και αυγά από κλωνοποιημένα ζώα, ακόμα και αν η FDA λέει πως αυτά είναι ασφαλή. Επίσης επιμένουν ε, το 89% των Αμερικανών καταναλωτών θέλουν να φέρουν ετικέτες ε, τα προϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα, ενώ 46% έχουν ηθικές ε, αντιρρήσεις. πόσο εκτεταμένη είναι η ε, κλωνοποίηση των ε, ζώων των ζώων. Δεν υπάρχει εμπορική κλωνοποίηση ζωντανών ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχουν ε, σχέδια για να χρησιμοποιηθεί πριν το 2020. Η εμπορική κλωνοποίηση επικεντρώνεται στι ΗΠΑ, στον Καναδά και την Αργεντινή. Επίσης υπάρχουν κάποιε δραστηριότητε στη Νέα Ζηλανδία, στην Αυστραλία, τη Χιλή, την Κίνα και κάποιες νοτιοαμερικανικέ χώρε. Ε, ε, ε, εφαρμόζεται περισσότερο στο, στα βοηδή αλλά και στα γαλακτοπαραγωγικά ζώα. Επίσης στα χοιρινά στην Κίνα, και στην Κίνα όμως η κλωνοποίηση για τα εγωπρόβατα δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Τώρα, η χνηλασιμότητα. Οι περισσότερες τέτοιες χώρες δεν ρυθμίζουν τα τρόφιμα από κλωνοποίηση με το μόνο εξαίρεση τον Καναδά που θεωρεί ότι το τρόφιμα από κλώνους και τα απογόνους ε, και νέα τρόφιμα και απαιτεί ε, αξιολόγηση ασφάλειας πριν αυτά να τεθούν σε εμπορία. Ε, επίσης σε κάποιες τέτοιες χώρες, όπως στην Αυστραλία, υπάρχει θελοντική σήμανση Εν γέννη τι χώρες πάντως δεν διακρίνουν ανάμεσα στου κλόνου και τα παραδοσιακά ε, ζώα. Ε, υπάρχει ωστόσο κάποια εξαίρεση στη Νέα Ζηλανδία όπου υπάρχει σύστημα εντοπισμού και ιχνηλασιμότητα, και αυτό με στόχο τι ξένε αγορέ κυρίως. Υπάρχουν επίσης ιδιωτικέ πρωτοβουλίε στον Καναδά, τη ΣΥΠΑ και τη Βραζιλία όπου ορισμένε χώρε ε, κρατούν όπου αυτές οι χώρες μάλλον ε, ε, κρατούν ε, μητρώα για τους κλόνους. Στην Ένωση έχουμε ήδη την ταυτότητα για, για το σπέρμα αλλά και για τα έμβρια. Αλλά δεν ξέρουμε αν αυτά προέρχονται από κλωνοποιημένο δότη. Υπάρχουν επίσης κάποιες συμφωνίες ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Καναδά που επιτρέπουν τον εντοπισμό υλικού αναπαραγωγικού υλικού από Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντωμεταξύ έχουμε ειχνηλασιμότητα για τα, ε, για το, το βόλιο κρέας, για τα εγωπρόβατα, αλλά και χνηλασιμότητα για τα χείρου. Ε, ενώ στην ε, ΣΥΠΑ όχι. Εδώ έχουμε ένα πίνακα, φαντάζομαι δεν το βλέπετε πολύ καλά, πάντως ε, πρόκειται για μια μαρτυρία που δόθηκε στο ε, Αμερικανικό Υπουργείο, ε, στο Αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας από τον ανώτατο πολιτικό αναλυτή για την κλωνοποίηση και τα γενετικά τροποποιημένα ζώα είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρξει εντοπισμός της κλωνοποίησης στην καταγωγή του ζώου. Δυστυχώ αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στην πρόταση του εις Κομισιόν του Δεκεμβρίου 2013. Ε, σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τρόφιμα από κλόνους θεωρούνται νέα τρόφιμα και άρα χρειάζεται έγκριση πριν να τεθεί σε εμπορία. Ε, όμως δεν ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες για τα τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα. Πριν από μερικά χρόνια, το 2010, στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκαλύφθηκε ότι τρόφιμα, ε, ε, δηλαδή κρέας και γάλα, είχαν μπει στην διατροφική αλυσίδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν υπήρχε τίποτα παράνομο, αλλά ήταν σοκαριστικό για τους Βρετανούς καταναλωτές ότι δεν μπορούσε κανείς να πει αν έτρωγε ε, τρόφιμα από απογόνους κλώνων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και αντίθετα με τη μικρή γελιογραφία που βλέπετε κάτω αριστερά στην διαφάνειά μου, θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι οι κλόνοι είναι παντού στην αγορά και ότι οι καταναλωτές ήδη καταναλώνουν κλωνοποιημένα προϊόντα. Η κλωνοποίηση είναι νέα τεχνική, το ποσοστό επιτυχία είναι πολύ χαμηλό και γι' αυτό έχουμε χρόνο, αν θέλουμε να το κάνουμε, να ρυθμίσουμε νομοθετικά την κλωνοποίηση ζώων για την τροφική αλυσίδα και έχασε μια ευκαιρία η Κομισιόν γιατί θα μείνει ε, ναι, ο καταναλωτή στο σκοτάδι όσον αφορά ε, του απόγόνου κλώνων. Είναι υποκριτικό να απαγορεύουμε κλώνους και τρόφιμα από κλώνου όταν ξέρουμε πω οι κλώνοι κατασκευάζονται για, λόγους, ε, για σκοπούς αναπαραγωγής ενώ οι απόγονοι για την παραγωγή γάλακτος κυρίως. Εδώ έχουμε κάποιες εμπορικές πτυχές ε, ε, όσον αφορά ε, τη νομοθεσία που μπορεί να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ πάλι το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επιτρέψει τη χρήση κλωνοποιημένων ζώων ή προϊόντων από τους ε, απογόνους. Γι' αυτό υπάρχει χρόνος να ρυθμίσουμε νομικά τα θέματα. Η Κομισιόν θέλει να προχωρήσει περισσότερο και να προτείνει απαγόρευση της εισαγωγής ζώων των κλώνων στην ε, ευρωπαϊκή αγορά. Όμως δεν κάνει τίποτα όσον αφορά το ε, αναπαραγωγικό υλικό. Εμείς συμφωνούμε με τους εμπορικούς εταίρους της Ένωσης ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να αλλάξουμε το τελικό περιεχόμενο της πρότασης της Κομισιόν. Έχουμε εδώ δηλώσεις από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη ΣΥΠΑ, όπου σαφώς εστάλει μήνυμα στην Ένωση πως οι χώρες αυτές θα παρακολουθούν πολύ στενά τις συζητήσεις για το θέμα αυτό στην Ένωση και θα ήθελαν οποιοδήποτε κανονισμός να παραμείνει αυστηρά στην, στα επιστημονικά δεδομένα. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις διαπραγματεύσεις με, για το, την ΣΕΤΑ και την ΤΙΤΙΠ. Οπότε δεν μπορούμε παρά να προβληματιζόμαστε όσον αφορά την επιρροή που ασκούν αυτές οι διαπραγματεύσεις εμπορικές στις προτάσει προτάσεις της Κομισιόν. Άρα λοιπόν τελικά θα πρέπει να πούμε ότι ο καταναλωτή θα πρέπει να είναι ενήμερο όταν θέλει να αγοράσει και να καταναλώσει τρόφιμα που προέρχονται από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων. Τουλάχιστον θα θέλαμε να δούμε απαγόρευση κλωνοποίηση των ζώων για παραγωγή τροφίμων επίσης απαγόρευση των τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα και των εισαγωγών των κλώνων για παραγωγή ε, τροφίμων. Αυτό ήδη υπάρχει στην πρόταση της Κομισιόν και με αυτό συμφωνούμε. Θα θέλαμε επίσης συχνηλασιμότητα για το ε, σπέρμα και τα έμβρια κλωνοποιημένων ζώων, αλλά και για τα ζωτα... τους ζωντανούς απόγονους κλωνοποιημένων ζώων. Βασικά αυτό ε, σχεδόν συμφώνησαν επ' αυτού μάλλον το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από τρία χρόνια και πιστεύουν πως ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Βεβαίω θα θέλαμε όλα τα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και από γόνους αυτών να φέρουν συγκεκριμένη σήμανση. Ξέρουμε ότι είναι αυτό υποσυζήτηση. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό η πίεση από τους εμπορικούς εταίρους των, των, της Ένωσης να μην εμποδίσει την Ένωση ε, να υιοθετήσει κανόνες ε, που είναι σύμμορφοι προς τα αιτήματα των πολιτών. Το 2011 διέρευσε μια γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου που έδειχνε πως οι απαιτήσει σήμανσης για τα τρόφιμα και για τα ζώα από μάλλον τα τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα και αποχώνους δεν ήταν συμβατή με τις απαιτήσεις του ΠΟΕ και της ΓΚΑΤ. Περισσότερο από εμπόδιο πιστεύουμε ότι η διαπραγματεύσει με την ΤΥΠΗ θα ήταν μια ευκαιρία για την Ένωση και τη ΣΥΠΑ να υιοθετήσουν κανόνε για την κλωνοποίηση των ζώων προ το συμφέρον των καταναλωτών. Άκουσα νωρίτερα πω ίσω οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ να έχουν μια ιδιαίτερη στάση απέναντι στη τεχνολογία και την κλωνοποίηση. Πάντω, μαζί με του ε, ομολόγου μα ε, τη Αμερική, εμεί εκπονήσαμε ένα ψήφισμα που έχει φέρει τον τίτλο TACD και θα δείτε ότι έχουμε παρόμοια αιτήματα με τους ομορικανούς ομολόγους μας. Καλωσορίζω λοιπόν το πρόσκλησή σας να... και την διάθεσή σας να ακούσετε τη γνώμη των καταναλωτών και προσβλέπω στις επόμενες συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Περνάμε στη συζήτηση. Το λόγο έχει ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ομιλητές. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία που ανέφεραν και αφορούν κάπως την, περι... την ε, Επιτροπή ΕΝΒΗ. Πρώτα απ' όλα η συζήτηση με τους υπόλοιπους ε, εταίρους μας πράγματι από ό,τι φαίνεται ο Επίτροπος Μπόρκ πήγε με μια πιο φιλόδοξη πρόταση εντός της Κομισιόν και οι υπόλοιποι επίτροποι τον εμπόδισαν ε, με το επιχείρημα μεταξύ άλλων πώς θα διακινδυνεύσουν οι εμπορικές σχέσεις με τη ΣΥΠΑ. Εγώ είμαι υπέρ της συμφωνίας TTIP αλλά το είπε ήδη η Κομισιόν τους είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στον κόσμο το ότι δεν προτείνουμε καν πλέον νομοθεσία γιατί δεν θα αρέσει στους Αμερικάνους. Ε, Κάπω κάπως αλλιώς πρέπει να κάνουμε τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα να ε, πούμε τι θέμε εμείς και μετά να διαπραγματευτούμε. Και ας γίνει ένα συμβιβασμός. Αλλά δεν θα το δεχτεί κάτι τέτοιο το κοινοβούλιο, το να μην υπάρχει καθόλου πρόταση. Δεύτερον, η δυσκολίες με τη σήμανση. Ομολογουμένως δεν είναι κάτι το απλό, αλλά πρώτα απ' όλα ε, εμένα η πτυχιακή μου εργασία αφορούσε την ε, γενετική και την διάγνωση in vitro και πήγα και σε μια συγκεκριμένη εταιρεία που παρασκευάζει ακριβώς ε, τέτοιο υλικό και κάνει τέτοιες δοκιμές. Και τους ρώτησα, εάν εμείς αποφασίσουμε πώς α, ε, θέλουμε να υπάρχει σήμανση του κρέατος που προέρχεται από τέτοια ζώα, μπορείτε να μας φτιάξετε ένα τεστ έτοιμο και μας λέει ναι δώστε μας μερικούς μήνες και θα το έχουμε. Οπότε τώρα μιλάμε για, για τρόφιμα Ε, πρόκειται για πράγματα τα οποία έχουν μέσα τους και DNA έτσι. Οπότε το θέμα είναι ποιος μας δίνει ακριβώς τις γενετικές πληροφορίες για τα κλωνοποιημένα ζώα. Υπάρχουν κάποιες ε, χιλιάδες ε, ζώα από τα οποία προέρχονται όλα τα υπόλοιπα. Ακούσαμε ήδη και στη συμβατική γεωργία από ένα ζώο καταλήγουμε να έχουμε 500.000 απογόνους. Όταν λοιπόν αγοράζουμε σπέρμα ή ένα έμβριο με πολύ υψηλή τιμή γιατί μας ε, λέει ο παραγωγός ε, ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό ζώο, δεν είναι δυνατόν μετά να μας λέει ότι δεν ξέρω αν εκλονοποιημένο ή όχι. Αν πληρώνω εγώ γιατί αγοράζω καλό γενετικό υλικό, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να εξετάσουμε εάν πραγματικά είναι από το συγκεκριμένο ζώο ή από κλωνοποίηση. Λίγη καλή θέληση χρειάζεται, δεν μπορεί να μας λέτε ότι δεν γίνεται και αυτή η καλή βούληση θα βρεθεί και στις ΗΠΑ και στις λατινοαμερικάνικες χώρες αν επιδείξουμε και εμείς λίγη πολιτική βούληση. Δεν μπορεί κανείς ε, να με πείσει ως επιστήμονα από αυτά τα οποία ξέρω πως είναι αδύνατον κάτι τέτοιο. Έχουμε ήδη κανόνες ε, που ισχύουν που λένε πως η προέλευση του νοπού κρέατος και στο χείριο και στα πουλερικά θα πρέπει να γνωστοποιείται. Αυτό δεν γίνεται με DNA, χρειάζεται απλά να δοθούν οι πληροφορίες. Και έτσι νομίζω θα αναγράφονται και πληροφορίες για την ε, γενετική προέλευση των ζώων. Τελευταίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ομάδας για την ε, δεοντολογία. Γιατί είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι όσο πιο καλά πάει η τεχνολογία στα ζώα, τόσο πιο γρήγορα θα μεταφερθεί στους ανθρώπους. Και ευτυχώς από ό,τι φαίνεται το επιχείρημα που έχω ακούσει είναι ότι δεν θα γίνει αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλές βλάβες ε, στα, στα ζώα και ό,τι γίνεται στα κλωοποιημένα ζώα θα γίνει και με τους ανθρώπους. Οπότε, αν κλωνοποιηθεί η κλωνοποίηση των θηλαστικών έτσι ώστε να μην υπάρχουν πλέον προβλήματα. Κάποιοι ε, επιστήμονες, δεν ξέρω ποιοι θα είναι και πού θα είναι, γρήγορα θα πούνε «Ε, «Εντάξει, άμα γίνεται στα ζώα, μπορεί να γίνει και στον άνθρωπο» χωρίς ε, παρενέργειες. Και αυτό νομίζω από μόνο του είναι ε, σημαντικό επιχείρημα. είναι νομίζω σαφές πως είμαστε κατά μιας τέτοιας εξέλιξης, ε, γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να το εμποδίσουμε από τώρα. Όταν λένε οι επιστήμονες πως ε, με τα χρόνια τα ζώα δεν θα υποφέρουν, είναι μια επικίνδυνη συζήτηση στην οποία ε, μπαίνουμε, γιατί όλο και κάποιος θα πει ας το δοκιμάσουμε και στους ανθρώπους. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Thank ευχαριστώ. Κυρία Μιούλερ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, και εγώ έχω ερωτήσει για την ΕΦΣΑ. Υπάρχουν εκτιμήσεις για τις ποσότητες των εισαγόμενων τροφίμων που προέρχονται από κλόνους. Και όταν μιλάμε για εισαγωγές από ΙΠΑ, μήπως πρόκειται για τρόφιμα τα οποία θα έπρεπε να έχουν ειδική άδεια. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των κλώνων είναι κάπως πιο ασθενές. Ε, αυτό αφορά νομίζω και τους απογόνους τους και θεωρώ πως ο, ο που είπε εδώ πέρα πως ε, θα πρέπει να υπάρξει μια ανάλυση του DNA. Δεν έχω πιστεί ακριβώς γιατί όταν έχουμε το σπέρμα ενός ε, τάβρου και μετά είναι του κλωνοποιημένου ζώου ακριβώς το ίδιο, θα είναι ίδιο και το DNA. Το να συμπεράνουμε λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε τη διάκριση, δεν ξέρω από πού βγήκε. Ε, θα ήθελα μια απάντηση από εσάς. Και τέλος, εάν πράγματι ε, είναι ασθενέστερο το ανοσοποιητικό τους, τι σημαίνει αυτό για την διατροφική μας ασφάλεια. είναι κάτι το οποίο θα ξέρουμε, πως είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Γιούζο. Ευχαριστώ. Έχω ένα σχόλιο και μία ερώτηση προς τον κύριο ε, Πέρε Πουικτομένετς. Μιλήσετε για προβλήματα διοντολογίας, ε, προβληματισμός προς την ευημερία των ζώων, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι αν θέλουμε να αντιταχθούμε στην κλωνοποίηση, αυτά τα επιχειρήματα θα πρέπει να προτάξουμε. Επίσης, για το θέμα της επιστηστικής ασφάλειας, ε, σε πολλές τις εκθέσεις ε, η ΕΦΣΑ δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το κρέας ή το γάλα ενός κλωνοποιημένου ζώου ή του απογόνου, του, του απογόνου τους δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Βέβαια το κρέας του κλωνοποιημένου ζώου του ίδιου δεν καταναλώνεται. Των απογόνων κυρίως καταναλώνεται. Προσοχή όμως, μήπως πέσουμε στην ίδια μας την παγίδα. Σε ό,τι αφορά την πολυμορφία, τη γενετική. Όταν κλωνοποιούμε ένα ζώο δεν κάνουμε γενετική μετάλλαξη όπως γίνεται με τους σπόρους. Κλωνοποιούμε ένα και μόνο ζώο την ίδια επιλογή την κάνουμε και χωρίς κλωνοποίηση. Οπότε διαφωνώ. Αυτό γινόταν ανέκαθεν και στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Γίνεται επιλογή για την αναπαραγωγή ε, τα καλύτερα άτομα. Το χρησιμοποιούμε ε, επειδή έχει καλύτερα, τα καλύτερα χαρακτηριστικά. Ε, και στην ε, Ισπανία είχαμε ένα τέτοιο, μια κλοποίηση ενός πολύ ποιοτικού τάβρου και δεν έχω, δεν έχω καμία αφιβολία ότι τα προϊόντα των απογόνων δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα στην κατανάλωση. Δεν υπάρχουν προβλήματα επιστήστικης ασφάλειας. Υπάρχουν διοντολογικά προβλήματα και προβλήματα ευημερία ζώων. Αυτό θα πρέπει ε, να θέσουμε ως επιχείρημα. Θέλουμε να αντιταχθούμε στην κλωνοποίηση. Όχι όμως στην επιστήστικη ασφάλεια, γιατί με αυτήν δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ. κύριε Αγγιλέρα. Ευχαριστώ. Έχω πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Τη μία την έθεσε και με πρόλαβε η κυρία Γιούσου. Τι γίνεται με, το, με υποτιθέμενο πρόβλημα της γενετικής πολυμορφίας. Εγώ δεν βλέπω πρόβλημα, θα ήθελα να μου το εξηγήσετε. Συμφωνώ με το επιχείρημα της κυρίας Αγιούσο, ότι αυτό έγινε, γινόταν ανέκαθεν στη Γεωργία, η επιλογή δηλαδή, και δεν επηρέασε καθόλου την πολυμορφία, όπως σωστά είπε η κυρία Γιούσο. Ε, η εκπρόσωπος της Οργάνωσης των Καταναλωτών θα ήθελα να μου πει το εξής, μια και μελέτησε πολύ διεξοδικά όλα αυτά τα θέματα. Πιστεύετε ότι όταν ρωτάτε τον κόσμο για την κλωνοποίηση γνωρίζει ο κόσμος τι, τι ακριβώς θα πει κλωνοποίηση ή ταυτίζει την κλωνοποίηση με τη γενετική μετάλλαξη, κάτι που είναι τελείως λάθος. Μήπως απλώς ο κόσμος ακούει κλωνοποίηση και επειδή έχει κάποια διοντολογικά προβλήματα προκαταλαμβάνεται και απαντά αρνητικά χωρίς όμως να γνωρίζει πραγματικά τι εστί κλωνοποίηση. Και λέω κάτι τέτοιο ότι μερικές φορές ακόμη και οι εμπειρογνώμονες δυσκολεύονται να καταλάβουν και γίνεται συχνά μια εκστρατεία υπέρ ή κατά κάποιου θέματος και μερικές φορές εσκεμμένα ε, ταυτίζουμε τη μετάλλαξη, την κλωνοποίηση με αρνητικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. Πιστεύετε ότι ο απλός καταναλωτής γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ κλωνοποίησης και γενετικής μετάλλαξης ή γνωρίζει τι σημαίνει πραγματικά κλωνοποίηση. Νομίζω είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, για να κρίνουμε πόσο ακριβείς είναι οι απαντήσεις που δόθηκαν. Επίσης, ε, θα ήθελα να δηλώσω και πάλι ότι έρευνα σημαίνει εξέλιξη και άρα πρόοδος. δεν πρόκειται ποτέ να αντιταχθώ στην έρευνα και την εξέλιξη. Φυσικά με επιφυλάξεις, με ασφαλιστικές δικλίδες. Όταν έγιναν έρευνες στην πατρίδα μου, στην Ισπανία και στην δική μου περιφέρεια για τα βλαστοκύτταρα και τη βελτίωση που θα επιφέρουν στην υγεία και στην ποιότητα ζωής, στην αρχή όταν μιλήσαμε για τα βλαστοκύτταρα ήταν πολύ κατά στην ε, ιατρική έρευνα. Αλλά ήταν σημαντικό το έργο που έγινε στα βραστοκύτταρα. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσει εδώ, αλλά σας λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μερικέ φορέ κάποια θέματα προβάλλονται με συγκεκριμένο τρόπο στην κοινή γνώμη για να προκαλέσουν θετική ή αρνητική αντίδραση. Παρά τις αρχικές αντιδράσεις είδαμε ότι η αρνητικη αντιδραση παρα τι αρχικέ αντιδράσει ειδαμε οτι η ερευνα στα βραστοκύτταρα θα αποφέρει καρπούς. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να κάνω εδώ συγκρίσει ή παραλληλισμού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αντιταχθώ στην έρευνα. Αλλά με εχέγγυα, με ασφαλιστικέ δικλείδε. Και συμφωνώ ότι εδώ έχουμε ε, κάποιες ανησυχίες ως προς την ε, ευημερία των ζώων. Εκεί υπάρχουν εύλογες ε, ανησυχίες για την ευημερία των ζώων και τις καλές συνθήκες διαβίωσης. Και αντιλαμβάνομαι και τα δεοντολογικά προβλήματα που σας έχουν μερικοί με την κλωνοποίηση. Και για την είσοδο στην αλυσίδα ε, των τροφίμων, στη διατροφική αλυσίδα, αλλά και για αυτά που είπε ο κύριος Λίζε. Αν, πολλοί φοβούνται ότι αν η κλωνοποίηση τελειοποιηθεί, πολλοί φοβούνται ότι θα περάσουμε και στην κλωνοποίηση ανθρώπων. Και εκεί είναι που πανικοβαλόμαστε όλοι. Υπάρχουν λοιπόν δεντολογικά προβλήματα, θέματα με την ε, ευημερία των ζώων, αυτά έχουν μείνει ανεπίλητα ακόμη. Θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη λοιπόν στις ε, πιθανές νομοθετικές ρυθμίσεις. Αλλά εδώ μιλούμε για οδηγία απαγόρευσης. Απαγόρευσης. Και πέραν κάποιων βελτιώσεων που θα πρέπει να γίνουν, κατά τη γνώμη μου το σημείο αφετηρίας της οδηγίας δεν είναι καθόλου κακό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρεκ. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προλαλήσαντες για αυτά τα οποία μας είπαν, πολύ ενημερωτικά και κατέδειξαν μία τάση. Εγώ όμως θα ήθελα να πω το εξής. Στην κοινωνία μας, όλο και περισσότερο, ε, αμφισβητείται η σχέση ανθρώπων ζώων στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Να, κυρίως στην Ευρώπη. Και άρα δεν είναι ε, να απορούμε για το ότι μία ε, ομιλήτρια είπε πως 66% των καταναλωτών, 66 των καταναλωτών ε, δεν θέλουν τα κλεινοποιημένα προϊόντα για λόγους δεοντολογίες. Να πω πως τα τελευταία 100-150 χρόνια το το ζώο έχει γίνει καθαρά ένας ε, παραγωγικός συντελεστής και τίθεται το ερώτημα τι άλλο θα κάνουμε στα ζώα. Και δεν νομίζω πως είναι η θέση μας να παίζουμε τον Θεό εδώ πέρα, να επεμβαίνουμε στην εξέλιξη και να κλωνοποιούμε ζώα. Κάποιοι λένε εντάξει η επιστημονική πρόοδος, αλλά ε, που μας έφερε η επιστημονική πρόοδος ο Αϊνστάιν όταν είδε το τι έκανε η βόμβα στην Χειροσύμα είπε πως έπρεπε να τα, τα αφήσουμε αυτά τα πράγματα ήσυχα τελικά. Δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει λοιπόν μια μέρα η κλωνοποίηση. Το οφείλουμε λοιπόν στους Ευρωπαίους καταναλωτές να υψώσουμε το αναστημά μας στην Αμερική και να πούμε Αφήστε το τώρα, άμα θέτε κλωνοποιημένο κρέας, φάτε το εσείς. Εμείς ε, θα συμπεριφερθούμε κάπως διαφορετικά και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού κάντε εσείς ό,τι γουστάρετε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόγκοβιτς έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ε, παρουσιάσεις σας μας βοηθούν πάρα πολύ σε αυτά τα περίπλοκα ζητήματα. Εγώ στηρίζω την άποψη όσων λένε πως ε, θα πρέπει να δούμε την πλευρά της ε, δεοντολογίας. Γιατί όταν μιλάμε για αμφισβήτηση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών το ίδιο και περισσότερο ε, ισχύει και για τους ε, κλόνους. Γι' αυτό εγώ προσωπικά είμαι στο πλευρό αυτών που είναι πολύ επιφυλακτικοί για το θέμα αυτό. Θεωρώ πως το θέμα της διοντολογίας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί Σήμερα απειλούμαστε κυρίως λόγω ζητημάτων οδεοντολογίας και ηθικής, όχι τόσο τεχνολογίας. Είμαστε στο έτος 2015 και συζητάμε και θα συζητήσουμε φέτος και για το TTIP. Και εγώ είμαι με αυτούς που θεωρούν πως θα πρέπει να τοποθετηθούμε σαφώς πριν από τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με τις ε, διατλαντικές ε, αυτές ε, διαπραγματεύσεις. Αυτά και συμφωνώ με αυτούς που έχουν κάποιες επιφυλάξεις ηθικής φύσεως. Σας ευχαριστώ, δεν βλέπω κάποιο αίτημα από τους βουλευτές. Δίνω λοιπόν αμέσως τον λόγο στους εμπειρογνώμονές μας με τη σειρά που μίλησαν και πριν. Ο κύριος Ρόμπινσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα ζητήματα που ετέθησαν στον τομέα του εμπορίου η λασιμότητας και όλα αυτά τα θέματα που είναι εκτός της αρμοδιότητάς μας ε, οπωσδήποτε δεν θα αναφερθώ θα τα αφήσω στους άλλους ομιλητές όσον αφορά τις εκτιμήσεις ε, των τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα δεν τα έχουμε δεν έχουμε τέτοια νούμερα το θέμα των εξασθενημένων ε, ανοσοποιητικών των κλωνοποιημένων ε, ζώων και των απογόνων τους. Βλέπουμε παρόμοια διάρκεια ζωής, παρόμοιο αναπαραγωγικό δυναμικό και έχουν ε, λειτουργικά ανασωπητικά στήματα Τέλος για την γενετική ποικιλία το ζήτημα που μας απευθύνθηκε ήταν το τι ε, επίπτωση έχουν στο περιβάλλον, όχι στα ίδια τα ζώα. Στο περιβάλλον λοιπόν δεν είδαμε επίπτωση πέρα από τα αναμενόμενα. Δηλαδή στον τομέα της κοινοτροφίας όσα ισχύουν και στα μη κλωνοποιημένα ζώα δηλαδή. Ευχαριστώ. κύριος Επειδή πολλές ερωτήσεις τέθηκαν στα ισπανικά, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω και εγώ ισπανικά. Αυτό που είπα για την επιστημιστική ασφάλεια και τις ανησυχίες της, ομάδας, ε, της Ευρωπαϊκής Ομάδας ε, για την ε, διοντολογία. Σας είπα ότι κάναμε διαβουλεύσεις και καταγράψαμε αυτήν την ανησυχία. Αλλά κατά τη γνώμη μου, οι γνωμοδοτήσεις και της ΕΦΣΑ και της αντίστοιχης Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων μας καθησυχάζουν για την επιστημιστική ασφάλεια και τις συνέπειες των απογόνων κλωνοποιημένων ζώων στην ασφάλεια των τροφίμων. Οπότε δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ομάδα Διοντολογίας πρόβλημα με την επιστημιστική ασφάλεια, αλλά καταγράφουμε και λαμβάνουμε υπόψη τις καθησυχαστικές δηλώσεις της ΕΦΣΑ και της αντίστοιχης Αμερικανικής Υπηρεσίας τέθηκε υποθετικό κίνδυνο ως προς την επιστημιστική ασφάλεια και η ομάδα μας, η Ευρωπαϊκή Ομάδα Δεοντολογίας για την Επιστήμη και τις Νέες Τεχνολογίες ε, ε, θεωρεί ότι οι μεταγενέστερες ε, εκθέσεις δίνουν απάντηση καθησυχαστική σε αυτό το ερώτημα της ασφάλειας των τροφίμων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους πληθυσμούς κάποιων, κάποιων ρατσών ζώων, ε, σίγουρα ε, αυτοί οι πληθυσμοί είναι ακραίο παράδειγμα μείωσης. Μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα να είναι μόνο λίγα ζώα ε, η βάση για ολόκληρους γενετικούς πληθυσμούς. Γιατί αν διονύσουμε αυτό το μοντέλο, αυτή την πηγή και χρησιμοποιούμε αυτό το γενετικό υλικό πολλές φορές, ώστε δεν έχουμε από ένα τάβρο 500.000 απογόνους αλλά εκατομμύρια απογόνους, τότε όντως ε, μειώνεται η γενετική πολυμορφία, η ποικιλομορφία. Και αυτή την άποψη με τέτοια ε, μαζική χρήση συγκεκριμένου γενετικού υλικού υπάρχει πρόβλημα. Πάντως ε, αυτός ο τάβρο που κλωνοποιήθηκε τελικά δεν ήταν κατάλληλος και ε, εξαφανίστηκε γιατί δεν ήταν κατάλληλος για τευρομαχίες, ήταν δηλός Οπότε φαίνεται ότι το, η, η γενναιότητα δεν κληρονομείται με το DNA και όσο και αν αναπαράγουμε το DNA, τέτοια χαρακτηριστικά όπως τη γενναιότητα δεν μπορούμε να, την, ε, να τα αναπαράγουμε. Αυτό συνέβη με το συγκεκριμένο τάβρο της ταυρομαχίας που ο κλόνος του ήταν ακατάλληλος για ταυρομαχίες. Επίσης ε, δεν, μπορούμε, <laughs> δεν μπορείτε να περιμένετε από ένα επιστήμονα να πει ότι είναι κατά της έρευνας. Αλλά υπάρχουν ε, κάποιες εμπορικές διέξοδοι που οδηγούν σε αδιέξοδα και ίσως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά εξετάζουμε ένα θέμα που στα πλαίσια της γενετικής ε, τεχνολογίας και της εκτροφής είναι μάλλον δευτερεύον. Θα πρέπει επίσης να ακολουθήσουμε μία αναλογικότητα στις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Είναι σημαντικό. Γιατί μιλούμε για μικρό αριθμό ζώων. Και μιλούμε για περιθωριακή τεχνολογία. Όπως είπατε, η γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι είναι αυτοί που σε τελική ανάλυση θα αποφασίσουν τι θα χρησιμοποιήσουν στο αγρόκτημά τους και οι γεωργοί κτηνοτρόφοι δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την κλωνοποίηση. Ίσως χρησιμοποιηθούν, χρησιμοποιηθεί η κλωνοποίηση για άλλες εφαρμογές που είναι, ίσως είναι πιο ενδιαφέρουσες. Και υπάρχει και το θέμα της ανθρώπινης κλωνοποίησης που θα πρέπει να προσέξουμε. Um, Σας ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με το ερώτηση του κατά πόσο έχει ε, εισαχθεί στην Ένωση, έχουν εισαχθεί στην Ένωση τρόφιμα από τις ΗΠΑ, από που προέρχονται από κλόνους ή ε, από γόνους αυτών ε, και ε, δεν έχουμε καμία τέτοια, κανένα τέτοιο σχετικό στοιχείο. Αυτά τα κλωνοποιημένα προϊόντα, τα προϊόντα από κλωνοποιημένο υλικό έχουν θεωρηθεί νέα τρόφιμα και φέρουν σήμαση. Δεν νομίζουμε λοιπόν ότι έχει μπει στην ευρωπαϊκή αγορά ε, τρόφιμα από κλόνους ή από γόνους αυτών. Υπήρξαν ερωτήσεις ε, όπου προσπα... Ε, όσον αφορά την αξιολόγηση του κατά πόσο ο καταναλωτής μπορεί να διακρίνει τον κλόνο ή όχι. Ε, οι περισσότεροι μπορούσαν να πούν τι ακριβώς ε, συμβαίνει, αλλά όχι ακριβώς. Πάντως αυτό δεν έχει επηρεάσει τη θέση τους, γιατί οι ανησυχίες των καταναλωτών αφορούσαν, ε, μάλλον βασίζονται σε ηθικά ζητήματα. 77% των καταναλωτών θεωρούν ότι η, το κλωνοποίηση των ζώων μπορεί να οδηγήσει στην ε, κλωνοποίηση του ανθρώπου, για παράδειγμα. Και ότι ε, επίσης ε, μπορεί, υπάρχει ηθική αντίρρηση στην κλωνοποίηση. Θα πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν και για το στόχο όλων αυτών. Μιλάμε για τροφική αλυσίδα, για κατανάλωση σε τρόφιμα η αντίληψη είναι τελείως διαφορετική όταν μιλάμε για παραγωγή τροφίμων. Το χρειαζόμαστε την κλωνοποίηση για παραγωγή τροφίμων. Η απάντηση και η αντίληψη των καταναλωτών είναι πως όχι, δεν χρειαζόμαστε την κλωνοποίηση για αυτόν τον σκοπό. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα δίνω το λόγο στην Κομισιόν να μας εξηγήσει τη θέση της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Περισσότερο σχόλιο είναι, ε, γιατί θεωρώ πως αυτή η ακρόαση ε, είναι πολύ χρήσιμο πλαίσιο για να ορίσουμε τα προβλήματα που πρέπει να συζητηθούν. Καταρχήν αναφέρθηκε ότι θα έπρεπε να είναι δυνατόν να βρεθεί μία μέθοδος για να εντοπίσουμε ε, συγκεκριμένα τα ζώα όπου θα μπορούσαν να γίνει η κλωνοποίηση. Πάντως θεωρώ ότι αυτή, ε, μπορούμε ε, να βασιστούμε στο γενετικό υλικό. Αυτό που δεν μπορούμε να εντοπίσουμε είναι το αντίγραφο και το, ε, το αντίγραφο το κλωνοποιημένο ζώο και ο κλώνος του μπορούν να εντοπιστούν. Αν έχεις όμως σπέρμα δεν μπορείς να πεις αν είναι από το κανονικό ζώο ή από τον κλώνο του. Εκεί δεν μπορείς να πεις. Ε, αυτό σε σχέση με τα όσα είπα προηγουμένως ότι δεν έχουμε αντικειμενικό τρόπο να αναγνωρίσουμε το κλόνο από το πρωτότυπο. Δεύτερον, πιστεύω ότι όταν μιλάμε για την γενετική πολυμορφία, όντως ε, πρόκειται για μείωση της ε, γενετικής πολυμορφίας. Αλλά θα πρέπει να πω επίσης σαφώς ότι αν θέσουμε το ίδιο ερώτημα για την εντατική ε, γεωργία, πάλι θα πρέπει να απαντήσουμε ναι. Γιατί η εντατική γεωργία περιορίζει την γενετική πολυμορφία. Εξορισμού επιλέγουμε τα ζώα που δίνουν τα, αποτελέσματα, τα καλύτερα αποτελέσματα για τους δικούς μας στόχους. Και είτε δηλαδή θα πρέπει Μάλλον, ερώτηση δική μου είναι, θα σταματήσουμε τώρα την εντατική γεωργία, ε, τις εντατικές καλλιέργειες λόγω αυτού. Μάλλον όχι. Το θέμα είναι να δούμε ποιο τμήμα αυτής της γενικής τάσης ε, προκαλείται από αυτή την γενική τάση ή όχι. Ε, έπειτα, άλλο σχόλιο σχετίζεται με επανειλημμένα σχόλια τα οποία λένε ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα της κλωνοποίηση, γιατί μάλλον εξετάζουμε το θέμα της κλωνοποίηση επειδή να το ζητούν οι Αμερικανοί ή κάποιοι άλλοι. Εγώ θέλω να πω ξεκάθαρα ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να δεχτούμε ότι η κλωνοποίηση είναι ένα επιστημονικό αποτέλεσμα το οποίο έχει ε, αντίκτυπο και στην Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία του κοινού είναι κατά, υπάρχουν ε, άνθρωποι που πιστεύουν ότι έχει μεγάλο δυναμικό αυτή η τεχνολογία και στην Ευρώπη και αυτό ισχύει και για τους πρακτικούς και ότι αν δεν τα ρυθμίσουμε αυτά δεν θα έχουμε σαφείς κανόνες. Χρειάζεται ε, κανόνες στην Ευρώπη να υπάρχουν. Το κάνουμε αυτό για την Ευρώπη, όχι για τους Αμερικανούς. Πρέπει να βρούμε τις λύσεις μας ε, εδώ στην Ευρώπη και δεν αποτελεί αυτό απάντηση σε οποιοδήποτε αίτημα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ευρωπαϊκό θέμα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εδώ στην Ευρώπη. Τέλος, ε, με χαρά είδα ότι αποκρισταλώνεται τώρα, ότι έχουμε δηλαδή προβλήματα με την ευημερία των ζώων, έχουμε προβλήματα που σχετίζονται με, εθνικ... με ηθικές έννοιες και δεν έχουμε πραγματικά πρόβλημα με την ασφάλεια των τροφίμων. Ε, και ένας από τους λόγους που έχουμε... έχετε δύο προτάσεις και όχι μόνο μία είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη νομική βάση θα έλεγα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Ενώ για τα, την ευημερία του ζώων θα μπορούσαμε αυτό να το βασίσουμε σε συγκεκριμένα άρθρα. Για τις υπόλοιπες ε, σκέψεις είναι προβληματικό και γι' αυτό και αυτό το κομμάτι είναι χωριστό και χρειάζεται πραγματικά συζήτηση ε, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ηθικές ε, ανησυχίες. Πώς θα τις λύσουμε άλλο θέμα. Πάντως καταρχήν θα πρέπει να ακολουθήσουμε την νομοθεσία που ισχύει και τους κανόνες που έχουμε επιτάπητος. Και να πω επίσης ότι ενώ βλέπουμε και καταλαβαίνω τις ηθικές, τους ηθικούς προβληματισμούς που ξεπερνούν τα πλάτα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή αγαθών στην γεωργία ή στον τομέα της ε, γεωργίας. Όλα αυτά είναι ωραία και καλά, αλλά πρέπει να έχουμε ένα σαφή τρόπο για να δούμε πώς θα βασιστούμε και πώς θα προχωρήσουμε στην νομοθεσία μας. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Εμείς ευχαριστούμε. Και τώρα να δώσω και πάλι το λόγο στη συνεισηγητριές μας για τα τελικά του σχόλια. Πλέον κηρύξουμε το πέρα της πολύ αυτής ενδιαφέρουσας δημόσιας ακρόσεις. Πρώτα η κυρία Μόη. Σας ευχαριστώ. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ήδη μπόρεσα να πω στην αρχική μου ομιλία, ε, ακόμα έχω προβληματισμούς όσον αφορά την ανάλυση της ΕΦΣΑ για τη χρονοποίηση ε, τροφίμων. Θεωρώ πω είναι σύντομο το χρονικό διάστημα το το οποίο έγιναν οι μελέτε της ΕΦΣΑ. Πιστεύω πω η υγεία όλων των Ευρωπαίων πολιτών θα αξίζουν, αξίζει μεγαλύτερη προσοχή. Αρνούμε να πιστέψω πω η Ευρώπη θέλει να ασχοληθεί, ε, μάλλον θέλει να θεωρήσει ως πειραματόζα τους ίδιου του τους πολίτες, γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επιρροή στην υγεία των πολιτών ε, ε, από την κατανάλωση 20-30 ετών κλωνοποιημένων προϊόντων. 14 μήνε κράτησε η έρευνα και οι αναλύσει γίνανε στο εργαστήριο. Δηλαδή δεν έχουμε συγκεκριμένα και σίγουρα στοιχεία για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν δηλαδή στοιχεία. Μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υγείας στον πληθυσμό, τα οποία θα πρέπει να τα αναλάβει το δημόσιο σύστημα υγείας ε, το οποίο ε, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι σε θέση. Ε, τώρα, για τα ζώα, πιστεύω πως είναι καθήκον μας να μην δεχτούμε συμβιβασμού σε αυτό το θέμα. Το να εμποδίσουμε τα ζώα να υπόκειται σε ε, μαρτύρια θα πρέπει να είναι μία από τις αξίες που, τις μη διαπραγματεύσιμες που θα πρέπει να μας καθοδηγήσουν σε αυτή την πορεία. Θα πρέπει να, είμαστε, να διακρινόμεθα για την ποιότητα των προϊόντων μας ε, για να είμαστε ε, ανταγωνιστικοί δεν χρειάζεται να έχουμε ε, παραγωγή σε τεράστια κλίμακα, γιατί έτσι ε, ε, θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή των καταναλωτών μας. Έπειτα, πώς μπορούμε να εγγυηθούμε στους καταναλωτές μια εν γνώση τους επιλογή, μια ενήμερη επιλογή, όταν τα όσα ξέρουμε για, το, για την κλωνοποίηση είναι τόσο ευαίσθητα. Ξέρουμε, ας πούμε, πως τα κλωνοποιημένα ζώα δέχονται διάφορες αγωγές αγωγές με ορμόνες. Δεν ξέρουμε όμως ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτών των ορμονών στον άνθρωπο. Ε, βλέπουμε πως υπάρχουν ε, προβλήματα πνευμονικά, συστήματα ανοσοποιητικά, καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα. Θέλουμε αυτά να δούμε πόσο και κατά πόσο θα έχουν αυτά επιπτώσεις ε, στον άνθρωπο. Έπειτα, ε, η χνηλασιμότητα των ε, τροφίμων. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτε να γνωρίζουν τι βάζουν στο πιάτο τους. Ποιο μας εγγυάται πως ε, δεν χρησιμοποιούνται όλα αυτά για τα αγλοποιημένα προϊόντα για, για τροφικούς σκοπούς. Αυτό που αφισβητούμε δεν είναι η έρευνα. Πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στην κλωνοποίηση για ε, επιστημονικού λόγου και εκείνη που χρησιμοποιείται στη γεωργία και στην διατροφή. Θα πρέπει να αναζητήσουμε την επιστημονική βεβαιότητα. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβούν σφάλματα ε, από όπου δεν θα, μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα επιστροφή. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ υπεύθυνοι όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζόμερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. ήθελα να ευχαριστήσω και τους ομιλητές και τους ε, συναδέλφους ε, για τις ερωτήσεις τους. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε εν ολίγης πως οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι δεν το θένε. Δεν το χρειάζονται. Ο καταναλωτής δεν το θέλει. Και ακόμα και αν έχουμε τρόφιμα από απογόνους ε, τα οποία θεωρούνται με βάση τα σημερινά δεδομένα ασφαλή, ε, υπόθηκε πως δεν έχουμε μακροχρόνιες μελέτες. Ε, μετά έχουμε την προστασία των ζώων, υψηλή θνησιμότητα των ζώων και δυσμορφίες, επιπλοκές κτλ. κτλ. Μικρός, μικρό ποσοστό επιτυχίας, 6 μέχρι 15% στα βοηδή, 6% ε, μόνο στους χείρους. Ε, η διαδικασία υπάρχει ήδη 16 χρόνια και τα προβλήματα δεν έχουν μειωθεί Οπότε τα προβλήματα σε σχέση με τα ζώα, με τα ποσοστά θνησιμότητας ε, δεν λύνονται. Και από ό,τι φαίνεται οι προοπτικές είναι άσχημες ως ε, προς αυτό. Και δεν υπάρχει φως. Επίσης μιλήσατε για το τι γίνεται με οάρια και σπέρμα αποκλοποιημένες Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή η ίχνη λασιμότητα όταν μιλάμε για το πολλαπλασιαστικό υλικό. Και να πω πως υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν και στην ε, συμβατική γεωργία ε, βιβλία αναπαραγωγής ποιο ζώο ζευγαρώνει με ποιο, ε, πρέπει να είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο νομίζω και στην περίπτωση αυτή. Ναι, εντάξει, κοστίζει λίγο ε, παραπάνω, αλλά και στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς έχουμε ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας. Και εκεί πέρα δεν μπορεί, ε, και πράγματι δεν μπορούμε να αποδείξουμε στο εργαστήριο ότι ένα ζώο είναι κλωνοποιημένο, οπότε θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ειχνηλασιμότητας. Αυτό νομίζω προέκυψε από τη σημερινή συζήτηση. Κατόπιν. Υπάρχει η ανησυχία πως η μέθοδος αυτή θα χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους εάν επιτρέψουμε την ε, διάδοση της ε, κλωνοποίησης. αυτή τη στιγμή απαγορεύεται, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη και πώς θα μπορέσουμε να το εμποδίσουμε στο μέλλον. Από φαίνεται δεν έχει βελτιωθεί καθόλου η τεχνική θα γίνει δηλαδή σε περίπτωση που κλωνοποιήσουμε τη, γά, τη γάτα της γιαγιάς ας πούμε που πέθανε πριν από 60 χρόνια ή ένας συνάδελφος ανέφερε κάποια άλογα και εκεί πέρα ακριβώς όμως υπάρχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα, η υψηλή θνησιμότητα, δυσμορφία, η υψηλη θνησιμοτητα δυσμορφή, δυσπλασιες κτλ. δεν ναι, νομίζω να μπορέσουμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο αν το απαγορεύσουμε στα τρόφιμα. Πράγματι έχει πολύ σοβαρέ αντιρρήσει ή και είχε πολύ σοβαρέ αντιρρήσει στο Κοινοβούλιο. Τώρα θα δούμε. Δεν έχουμε τοποθετηθεί ακόμα στη νέα αυτή θητεία, αλλά προφανώ οι επιφυλάξει είναι οι ίδιε που είχε και ε, το προηγούμενο Κοινοβούλιο. Ναι, υπάρχουν ε, επιφυλάξεις όσον αφορά την προστασία των ζώων, όσον αφορά τα ζητήματα δεοντολογίας, και βέβαια όσον αφορά την ασφαλεία των τροφίμων. Και μετά μας λέτε πως πρόκειται για μια κάπως ε, περιθωριακή τεχνική. Ε, άμα είναι κάτι το περιθωριακό και δευτερεύον, είναι τόσο σημαντικό να το απαγορεύσουμε. Και αυτό τώρα έτσι μου ήρθε ως τελευταία σκέψη, αν είναι τόσο δευτερεύονται, δεν πειράζει και να το απαγορεύσουμε. Και τέλος... θα πρέπει να βρεθεί μια νομική ρύθμιση για το τι θα κάνουμε με τα ζώα εκείνα που προέκυψαν από την κλωνοποίηση δεν μπορεί να λέμε πως ε, εμείς απαγορεύουμε την κλωνοποίηση σε εμά και οτιδήποτε άλλο προκύπτει αλλού μπορεί να εισάγεται. Δεν ε, είναι δυνατόν. Έχουμε μία ευθύνη ε, και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, ναι, οι διαπραγματεύσεις του TTIP προχωράνε αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει ανεξάρτητη. Δεν χρειάζεται νομίζω πάρα πολύ ε, χρόνος, εάν το θέλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Αυτά και ευχαριστώ όλους όσους ε, συμμετείχαν. Θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε με το θέμα αυτό από εδώ και μπρος. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονές μας, τον Επίτροπο, τον μόνιμο αντιπρόσωπο της ε, Λατωνικής Προεδρίας και του συναδέλφους για την πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή συζήτηση που ήταν πολύ χρήσιμη για να κάνουμε περιστατωμένες ε, επιλογές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο τον κύριο Σικέρσκι για την πολύ επιτυχή διοργάνωση της δημόσιας Ακρός και την αγαστή συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκειά της. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα της συνεργασίας μας στο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε που και, και που θα είναι αναφυσβήτητα ιδιαίτερα καρποφόρο. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει αύριο στις 9 στην ίδια αίθουσα. Εδώ δηλαδή, ενώ η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει αύριο την τακτική συνεδρίαση στην 5G3. Οπότε λύεται η συνεδρίαση, αλλά πρώτα να δώσω το λόγο για μια σύντομη ανακοίνωση στο συμπρόεδρο τον κύριο Σικέρσικη. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη. Ε, οι κύριοι Ρεμπέκα και Ρίλκε σας προσκαλούν στην δημόσια ακρόαση για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της στρατηγικής ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημόσια αυτή ακρόαση θα γίνει σήμερα στην, σε 6,5 ώρα με συμμετοχή της Κόπα Κοζέκα και άλλων 5Β01. Απλώς θέλω να σας διαβιβάσω αυτό το αίτημα των δύο συναδέλφων. Ευχαριστώ. Λία τη συνεδρίαση.